Κυρίες και κύριοι, ε, συνήθως αρχίζουμε στην ώρα μας όταν εγώ προεδρεύω, ε, παρότι ο εισηγητής μας ο κύριος Λάιφρυντ ε, δεν είναι εδώ, ο κύριος Δεζίερ έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα κόλλημα, πρέπει να γυρίσει στη Γαλλία. Οπότε θα ρωτήσω, υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Uh, uh, Σημείο 6. Ε, αναβολή τη επόμενη συνεδρίαση στι 25 και 26 Οκτωβρίου. Σημείο 16, όχι 6 τη μέση διάταξη. Ήθελα να σα ενημερώσω. Κύριε Ντεζιρέ, ε, ζητήσατε αναβολή ε, ή θελήσατε να συζητηθεί νωρίτερα η έκθεσή σα, αλλά ίσω δεν είναι εδώ, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα είπαμε χθε το βράδυ, στείλαμε το μήνυμα σε 7.30. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, δεν ξέρω αν ε, το γνωρίζετε, γιατί είναι αρκετά σημαντική η έκθεσή σας. Αν δεν υπά... εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται η συζήτηση. Πολύ ωραία, εγκρίνεται η μέση διάταξη. Έγκριση των πρακτικών των της συνεδρίασης που έγινε στις 30 Αυγούστου του 2010. Θεωρώ τα πρακτικά εγκεκριμένα, εκτός αν προκύψει κάποιο άλλο θέμα μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, ανακοινώσει του Προέδρου σήμερα και αύριο αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίασή μας στο διαδίκτυο. Ε, έχουμε μοιράσει όλα τα έγγραφα που λάβαμε μέχρι σήμερα. Οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις απευθύνετε στη γραμματεία. Για το σημείο 22, δηλαδή ενδιάμεση συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη του Ειρηνικού. Θα έρθουν δύο υπουργοί από την Παππούα Νέα Γουινέα. Παππού Νέα Γουινέα. Ο Σάμιουελ Τ. Έιμπλ είναι υπουργό εξωτερικών εμπορίου και μετανάστευση τη Παππούα Νέα Γουινέα και ο κύριος Μπεν Σιμπράιτ, υπουργό Αλληλεία της Παππούα Νέα Γουινέα. Ε, επίσης, ε, πρέσβή ε, των Φίτζι, η εξοχότητά του, Βαν Βουικιού. μάλλον δεν πρόφερα σωστά το όνομά του. Στην έκτακτη συνεδρίαση ε, η έκτατη συνεδρίαση θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2010 από τις 9.30 μέχρι τις 10.30 για το Πακιστάν και ε, θα υποβάλουν αίτηση για το ε, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων Plus. Για το 2011 τώρα, η επόμενη συνεδριάση έχετε το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, ίσονος σημασία Εν γέννη, νομίζω, γίνεται εκτό το χρονοδιάγραμμα στη συνεδρία των συντονιστών. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Ωραία. Επιβεβαίνω τη έγκριση λοιπόν του χρονοδιαγράμματος. Σημείο 5. Τροποποίηση του κανονισμού περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης. Έχετε όλοι αντίγραφα. Um, Παρακαλώ, ε, Γιώργ, θα μπορούσες να μας ενημερώσεις ε, για την έκθεσή σου. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προκείμενη έκθεση είναι μια έκθεση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται σε ένα σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτό και αφορά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται διπλά για πολιτική χρήση και για στοχιωτική χρήση. Και εννοείται ότι το όλο θέμα συνδέεται και με ένα συγκεκριμένο βαθμό, αν θέλετε, ευαισθησίας. Από πλευράς περιεχομένου και μόνο, θα πρέπει να πούμε ότι η έκθεση αυτή προκύπτει από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εμείς ε, ως Επιτροπή την εξετάσαμε την πρόταση αυτή και υποβάλαμε και εκ νέου πρόταση για κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι σημαντικές προφανώς. να εξηγήσω κάποια από τις τροπολογίες αυτές και να πω και κάποια θέματα για το βασικό πρόβλημα της τροπολογίας, της ε, εκτασής αυτής. Θέλαμε να χρησιμοποιηθούν ε, οι διατυπώσεις από τις συνθήκες της Λισαβόνας και νομίζω ότι αυτό είναι δικαιολογημένο και θεωρούμε ότι στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να υπάρχει και μία συνάφεια, μία εναρμόνιση με άλλες ε, στοχοθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει φυσικά να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί ακριβώς αυτό επιτάσσει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Κάποια προβλήματα, λεπτομέρειες, τα οποία μπορούν να διευκρινιστούν Για να υπάρχει δηλαδή πιο πολύ έλεγχο επί τη αρχή για τι εμπορικέ αυτέ συναλλαγέ, να μην υπάρχει διαφορά σε ό,τι αφορά τον έλεγχο μεταξύ των κρατών μελών, να υπάρχει μια διέρεση, αν θέλετε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών, να υπάρχει και ένα κεντρικό έλεγχο στον τομέα αυτό. Μια άλλη λεπτομέρεια η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι το ερώτημα του πώς θα πρέπει να διεξάγονται οι τελικοί έλεγχοι γιατί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ένας έλεγχος της τελικής χρήσης. Επί της αρχής μπορούμε να πούμε ότι αυτό ασφαλώς ε, αποτελεί μια λύση, αλλά φυσικά συνεπάγεται και κάποιο άχθος, κάποιο κόστος. Από την άλλη πλευρά, ίσως θα μπορούσε να γίνει έλεγχος των τελικών χρηστών μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό επί της αρχής. Πώς τελικά δηλαδή θα πρέπει να διαμορφωθεί η πλέον κατάλληλη λύση και φυσικά να ακούσουμε και άλλες ε, απόψεις. Τώρα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ε, αναφοράς. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της πρότασής μας και της, προτασίας, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ένας έλεγχος, ε, μια υποχρέωση αναφοράς. χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά με μια έκθεση εξάντε. Ένα άλλο θέμα. Τι κάνουμε με τα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθέση. τα οποία ασφαλώς είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά πρινικά εργοστάσια. Όλα αυτά ασφαλώς θα μπορούσαν να συνεπάγονται κάποια προβλήματα. Είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό θεωρώ και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν σχετικές ρυθμίσεις. Και επίσης σε ό,τι αφορά τον κατάλογο με τις χώρες έχουμε κάνει κάποιες ε, ε, αν θέλετε, πολύ μικρές αλλαγές για να υπάρξει μια διαφορετική συστηματική, αλλά τα συζητάμε όλα αυτά. Τώρα, για θέματα περιεχομένου. Αυτά μάλλον όπως το περιεχόμενο. Κάτι άλλο τώρα. Πιο περίπλοκο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, βασίζεται σε, μια, σε ένα κανονισμό του 2000 και γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές τα προσαρτήματα. Παράλληλα όμως το Συμβούλιο προετοιμάζει και τροπολογίες σε κείμενο του 2009. Η λύση η οποία αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε στο ενδιάμεσο αν θέλετε πλαίσιο είναι να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε στο νομικό πλαίσιο του 2009, αυτό όμως ως υπόθεση, ως εικασία. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας επιβεβαίωσε την υπόθεση αυτή και θα πρέπει να ομολογήσω ότι και οι συνάδελφοι θεωρούν ότι σκόπιμα θα ήταν να απορρίψουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να βασιστεί στην τρέχουσα, ισχύουσα νομοθεσία και να υποβάλει εκ νέου σχετική πρόταση σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να εργαστούμε σε συνάρτηση με όσα κάνει το Συμβούλιο για να διορθωθεί κάπως αυτή η κατάσταση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ούτε ενθουσιασμένος είμαι με την πρόταση αυτή, ούτε και την απορρίπτω. Αν αυτό θεωρεί η Επιτροπή, δεν μπορώ να πω ότι θα την εμποδίσω. Αλλά αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι όχι, καλύτερα να συνεχίσουμε με την τρέχουσα πρόταση και να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, είμαι ανοιχτός και προς αυτή τη λύση. Να ακούσουμε τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι από τις άλλες ομάδες. Είμαι ανοιχτός πάντως σε ό,τι αφορά την κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο να κάνω μια εισαγωγή και είμαι πραγματικά περίεργος να ακούσω τι θα έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Γιώργο Ντανιέλ. Äh, Αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο εισηγητή για την εισαγωγή αυτή που έκανε. Νομίζω ότι κυρίως εξήγησε πάρα πολύ καλά την διαθεσμική κατάσταση πως έχει, ποιες είναι οι τυπικές δυσκολίες και οι διαφορές ε, ότι ουσιαστικά Συμβούλιο και Κοινοβούλιο εργάζονται βάσει διαφορετικού εγγράφου και στο Κοινοβούλιο ουσιαστικά επεξεργαζόμαστε ένα πεπαλαιωμένο κείμενο ενώ το Συμβούλιο έχει ένα τρέχον, πιο μοντέρνο κείμενο. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά κατά πόσον θα έπρεπε να ε, επιστρέψουμε. Να επαναπέμψουμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει νέα πρόταση η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν, συγγνώμη, λέει ο μιλητής, να σκεφτούμε λοιπόν ε, την επόμενη εβδομάδα κάποια πράγματα επί του περιεχομένου. Ο συναδελφός μας εξήγησε ποια θέματα τον απασχολούν ιδιαίτερα. Επίσης, μας, μας απασχολούν κάποιες προθεσμίες, γιατί πολλές επιχειρήσεις μου ανέφεραν ότι το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία για τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους για να απαντήσει κατά πόσον επιτρέπεται ή μη η εξαγωγή ενός προϊόντος. Αυτό θα ήταν σκόπιμο. Θα ήθελα να υπάρχει μια τέτοια προθεσμία. 6-8 εβδομάδες, 3 μήνες. Να το συζητήσουμε, δεν λέω, αλλά να λεφθεί μια απόφαση. Αν ε, η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει, να προβλέπετε ότι αυτόματα εγκρίνεται ή αυτόματα απορρίπτεται η αίτηση αυτή γιατί βλέπουμε ότι κάποιες επιχειρήσεις περιμένουν μισό, ένα έτος να εγκριθεί ή μη το αίτημά τους και νομίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί κανένα στα συμφέροντα. Δεύτερο θέμα το οποίο με απασχολεί και να το κοιτάξουμε. Το θέμα της ε, προκαταρτικής ε, έγκρισης, το θέμα της υποχρέωσης αναφοράς θέματα τα οποία με τον κανονισμό ουσιαστικά δυσκολεύουν εξαιρετικά την εξάγωγη των προϊόντων αυτών. Και ενδεχομένως τελικά τα προϊόντα αυτά, μάλλον να εγκρίνονται προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητες χρήσης και προορίζονται για στρατιωτική χρήση και να παρεμποντίζονται ε, προϊόντα για πολιτική χρήση. Γι' αυτό λοιπόν σωστό θα ήταν να κοιτάξουμε το κείμενο και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι σωστές ρυθμίσεις. Για το διαδικαστικό τώρα. Στην Επιτροπή να δούμε τι υποστηρίζει η πλειοψηφία, να υποβάλουμε τροπολογίες, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμβιβασμούς σε διάφορα θέματα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε αυτό δεν είναι θέμα και στην Ολομέλεια να ψηφιστούν αυτές οι τροπολογίες και αν είναι δυνατόν από τεχνικής άποψης να μην υπάρξει τελική ψηφοφορία αλλά να αναπαιμφθεί ο φάκελος να δώσουμε δηλαδή από πλευράς περιεχομένου α, κάποιες κατευθυντήρες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άποψη του Κοινοβουλίου αλλά με την αναπομπή να ζητήσουμε νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εξυπνάδα να συμπεριλάβει τα θέματα αυτά που θα προτείνουμε. Άρα να τοποθετηθούμε επί του περιεχομένου ως κοινοβούλιο, να μην ε, βάλουμε στον πάγο το θέμα αυτό και να δώσουμε τις προτάσεις αυτές στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, <clears throat> thank you, Daniel. Ευχαριστώ. ο Βίλιαμ έχει το λόγο. Διάβασα με ενδιαφέρον ε, το ζήτημα αυτό, παρόλο που τα σχόλια του εισηγητή ήταν ε, ιδιαίτερα τεχνικά. Πάντως νομίζω ότι δείχνουν παρόλα αυτά τη διάσταση απόψεων που υπάρχει. Όχι ανάμεσα στο EFD και στο EPP, ε, αλλά και ε, του, ε, του προοδρεύοντα της πολιτικής ομάδας ECR, δηλαδή ο, ο εισηγητής χρησιμοποιεί τη λέξη κοινότητα και όχι ένωση. Κοιτάξτε, μάλλον ε, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ένωση. Ένωση σημαίνει πολιτική ένωση που εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και μεγάλο μέρος ε, των πολιτών της Ευρώπης. Και, ε, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δεχθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας. Γι' αυτό λέω ο εισηγητής, που όταν θα αναδιατυπώσει την... Ε, την έκθεση, ίσως θα μπορούσε να ξαναβάλει τη λέξη κοινότητα και να σβήσει κάθε αναφορά στην Ένωση. Βλέπω ότι κάποιοι γνέφουν καταφατικά, άρα ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντω θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο προ το κατά πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικά. Ε, <coughs> Ευχαριστώ, Βίλιαμ. Και εγώ δεν μίλησα για το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω πώ ήρθε αυτή η ερμηνεία. Να ζητήσουμε στην Επιτροπή να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παύλο Κατζότη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία όσον αφορά το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι άκρος τεχνικό. Είναι μια τεχνική, όπω βλέπετε και στι πρόταση, και περιορισμένη ω προ το εύρο τη. Το Κοινοβούλιο στο μέλλον θα έχει επανειλημμένα ευκαιρίε να επανέλθει στη συζήτηση του ζητήματο ε, ε του, του ελέγχου των εξαγωγών των προϊόντων διπλή χρήση ε, στην ε, πολιτική της Ένωσης, εμπορική πολιτική της Ένωσης ε, προτιθέμεθα να ε, προτείνουμε διάφορες δράσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Βεβαίως, τα περισσότερα από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από τον εισηγητή μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους. Όπως σας είπα, αυτή η πρόταση που έχει ξεκινήσει το 2008 θέλει να δημιουργήσει ε, κάποια περιορισμένη φύσεως μέτρα διευκόλυνσης ε, για την εξαγωγή των προϊόντων αυτών, όμως διαφυλάσσοντας ε, απόλυτα θα έλεγα και διασφαλίζοντας απόλυτα τον, ε, τον έλεγχο, το βασικό έλεγχο ε, των ε, ελέγχων αυτών. Όπως τα ξέρετε, αυτό το, αυτά τα προϊόντα είναι, αναφέρονται στο 13% των εξαγωγών. Είναι μικρό σημείο, μικρό μέρος δηλαδή των εξαγωγών μας και κυρίως αφορούν τομείς της βιομηχανίας μας όπου ε, είναι πολύ σημαντική η ανταγωνιστικότητα και η υψηλή τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε μεταρρυθμίζουν το σύστημα του ελέγχου των εξαγωγών τους και, μέρος, και ως μέρος της δικής αυτής ο πρόεδρος Ομπάμα έχει θέσει ως στόχο να διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια οι εξαγωγές από τη ΣΥΠΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να καταβληθεί και περαιτέρω προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να δούμε ε, τι θα γίνει ε, και από ρυθμιστική άποψη και από κανονιστική άποψη όσον αφορά δηλαδή τον έλεγχο των εξαγωγών αυτών. Βεβαίω, λαμβάνοντα υπόψη ε, όλε τι πτυχέ που συνδέονται με την ασφάλεια και που είναι ο λόγο για τον οποίο επιβάλλονται αυτοί οι έλεγχοι σε τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Γκαζότη. Βλέπω ότι υπάρχει και εκπρόσωπο της ε, βελική Προεδρία. Θέλετε να σχολιάσετε αυτό το οποίο είπε ο Ντάνιελ. Όχι, πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ. Ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ επί τη ουσία με αυτά που είπε ο συνάδελφο Κασπάρη. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Επί του περιεχομένου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκόπιμο να διευκρινιστεί το θέμα της προθεσμιών που θα αφορούν τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες, να καθοριστεί ποιες είναι οι συνέπειες όταν δεν απαντά εντό της προθεσμίας η αρμόδια υπηρεσία. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτόν. Ο συνάδελφος Ντάτμας ε, θέλει να ξαναμπεί το community, το κοινότητα, αντί της Ένωσης Union, νομίζω ότι αυτό θα είναι δύσκολο για δημοκρατικούς λόγους, γιατί αποφασίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία ότι μιλάμε για Ένωση, δεν είμαστε πλέον κοινότητα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα και αν θέλετε τη γνώμη μου, καλώς έχουν όσοι έχουν τα πράγματα. Ίσως φυσικά άλλοι να έχουν διαφορετική άποψη, η οποία και είναι και σεβαστή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με λυπεί το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν εξετάζεται το βασικό μας πρόβλημα, τη νομική πτυχή. Μπορούμε να συζητάμε τεχνικά θέματα και ασφαλώς και θα καταλήξουμε σε κάποια ε, λύση. Αλλά το νομικό θέμα παραμένει ανεπίλητο. Θεωρώ ότι έπρεπε να λάβει το λόγο και να το αναφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έκανε. Ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε όπως πρότεινε ο συνάδελφος Κασπάρη. Να το δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν και να ακολουθήσουμε ίσως αυτή τη λύση. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Οκτωβρίου. Έγκριση της έκθεσης προβλέπεται για τις 9 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, προχωρά. Πάμε λοιπόν στην έκθεση Κούτας. Έχουμε λοιπόν το George εδώ. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ανησυχίε ε, ε, για το ότι στο ψήφισμα αυτό ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, πρέπει να εκφράσει στο ζήτημα αυτό το οποίο αφορά τι απαραίτητε αριθμητικέ προσαρμογέ που προκύπτουν την πρόθεση των ΗΠΑ να ανακαλέσει ειδικέ υποχρεώσει σύμφωνα με, τον, με την ΠΟΕ σχετικά με υπηρεσίε τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Αυτό το, αυτή η δέσμευση αριθμητικών προσαρμογών που ε, αφορά ε, τις υπηρεσίες αυτές, ε, τεχνικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αποθήκευση κτλ. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΠΑ ΕΕ, πήρε την απόφαση αυτή να κλείσει ε, ε, τις υπηρεσίες αυτές τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων που σημαίνει ε, τεράστιες απώλειες και από μεριάς κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έγινε κάτι τέτοιο σύμφωνα με το άρθρο 21 της Γενικής ε, ε, Συμφωνίας των Εμπορικών Υπηρεσιών άρα είναι απόλυτα νόμιμη υποχρέωση αυτή. Οι αντισταθμιστικές αυτές υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έγιναν στα πλαίσια του άρθρου αυτού. Άρα είναι επίση νόμιμε. Οι κανόνε ε, τη ΠΟΕ έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την ε, ε, αποφυγή μονομερών κυρώσεων και εμπορικών πολέμων. Όμω θα ήθελα να τονίσω ότι αυτέ οι αντισταθμιστικέ υποχρεώσει ε, πρέπει, πρέπει να εξεταστούν από κοινού με το συγκεκριμένο τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των στοιχημάτων. Εγώ συναντήθηκα προσωπικά με του βασικού εκπροσώπου του κλάδου και με ενημέρωσαν για το ότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, που εμπλέκονται, κυρίω οι υπηρεσίε online, οι εταιρείε online έχασαν τεράστια ποσά μέσα σε μία νύχτα. Και ορισμένε επιχειρήσει ε, ισχυρίζονται ε, ότι δεν είχαν δίκαιη μεταχείριση και από τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό συνιστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πολύ συγκεκριμένα ε, τις, ε, τα αιτήματα και τι προσφυγέ του κλάδου και να εξασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού ένα, ένα επίπεδο ισότιμη ε, μεταχείριση. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριε Κιούτα. Κύριε Γιακολίνο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και πιστεύω και εγώ ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ξεπερνά ε, την φύση του των διατάξεων που βρίσκονται υπό εξέταση. Και μάλιστα σας λέω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, εδώ αυτή τη στιγμή ε, ο Επίτροπο Μπαρνές εξετάζει ένα ευρύτερο έγγραφο το οποίο θα πρέπει να καθορίζει με ενιαία νομοθετική προσέγγιση το ζήτημα των τυχερών παιχνιδιών ε, στα, ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον εκ μέρου του κλάδου, όπως είπε και πολύ σωστά και ο, και ο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ε, τακτική των ΗΠΑ και τη κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν είναι πάντα ε, επικοδομητική ω προ τη συνεργασία. Βεβαίω θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη και οι ίδιε οι επιχειρήσει του κλάδου που θα πρέπει ε, που θα πρέπει να συμβάλλουν προς την εξυγίανση του κλάδου και να λαμβάνεται υπόψη το σύστημα των αδειών, εγκρίσεων κτλ. Τελειώνω αυτή τη σύντομη μου παρέμβαση και θα ήθελα ότι, να σας πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις πτυχές ε, των τυχερών παιχνιδιών και από την άποψη της υγείας αν θέλετε. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί και αυτή η πτυχή όταν μιλάμε για τα τυχερά παιχνίδια. Είμαι πεπισμένο ότι με τον συνάδελφο Κούτα και του άλλου σκιώδει συζητητέ και την Επιτροπή θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ευθύ αμέσω για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ορθολογικό ε, σύστημα το οποίο να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και που όπω σα είπα πριν από λίγο ε, είναι κάτι ή αποτελεί ένα αίτημα των εκπροσώπων του κλάδου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και εγώ είμαι σκιώδη και είμαι στον κατάλογο. Συμφωνώ με του προλαλήσαντε, με τον κύριο Κιούτο και τον κύριο Γιακολίνο. Πασκάλ Λαμή και ο ΠΟΕ εξετάζουν εκ του σύναγκη το θέμα. Συζήτησα με τον Πασκάλ Λαμή πριν από ένα δίμηνο για το αμερικανικό ζήτημα ε, και σίγουρα είχε επίγνωση όλων αυτών ε, Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που δεν του δίνουμε και πολύ σημασία γιατί θεωρούμε ότι τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια είναι κάπως ε, παράνομη δραστηριότητα από κάποιες ε, ε, πτυχές. Εντάξει, για τα περί υγείας συμφωνώ και ανησυχούν πολλοί άνθρωποι για αυτό το θέμα. Συμφωνώ με τον κύριο Κίουτα και τον κύριο Γιακολίνο. Θα ακούσουμε την Σάντρα Κάλχαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Καλημέρα σε όλους. Αντικαθιστώ τον ε, κύριο Γκάλαχαν, είναι συνάδελφός μου, Πολύν Βάντσιολ λέγομαι εγώ, είμαι από το ίδιο τμήμα στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου. Ασχολούμαστε με τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις και είμαστε επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων αυτών. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τον κύριο Γιακολίνο για τις παρατηρήσεις ε, που έκαναν. Πρώτη φορά εξετάζει η Επιτροπή το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω κάποια ζητήματα. Να σας δώσω και το υπόβαθρο. Υπάρχουν σοβαρότατες ανησυχίες για τα τυχερά παιχνίδια και λυπούμεθα που διαπιστώνουμε ότι η ΕΠΑ ε, υποχώρησε ως προς τις δεσμεύσεις της ε, στον κλάδο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο κλάδος ε, και είναι ισχυρότατη η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Άλλο ένα καθήκον μας, ε, θα, ε, μάλλον άλλο ένα θέμα είναι η συγκατάθεση που θα πρέπει να δώσει το Κοινοβούλιο μετά τη, το πέρας των διαπραγματεύσεων από το Συμβούλιο. Οπότε χαιρόμαστε που ενδιαφέρεται το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Council, um, decision, um, και αναμένουμε πρόοδο στη συζήτηση αυτού του ζητήματος. Ε, το πακέτο αποζημιώσεων αντισταθμίσεων ε, του 2007 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ ε, είναι καλό κατά τη γνώμη μας και δεδομένων των περιορισμών που έχουμε, ο εισηγητής συνόψισε με εξαιρετικό τρόπο την κατάσταση. Δηλαδή, είπα, υπαναχώρησαν από όλες τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει πρωτήτερα στον τομέα αυτό. Οπότε δεν υπάρχει ε, ένδικο μέσο για να ζητήσουμε αποζημιώσεις για τον άμεσα πληγέντα τομέα, δηλαδή του κλάδου των ε, τυχερών παιχνιδιών. Παρόλα αυτά, διαπραγματευτήκαμε, όπως έλεγα, ένα πολύ καλό πακέτο με τη ΣΥΠΑ και ας μην ξεχνούμε ότι ε, έχουμε καταλήξει νέες δεσμεύσεις σε βάση της Γενικής Συμφωνίας ε, Εμπορίου και Υπηρεσιών, το GATS δηλαδή, για τομείς κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τους courier, για τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, τις τεχνικές δοκιμές αποθήκευσης, Ξέρουμε ότι φυσικά αυτό δεν αντισταθμίζει τα τυχερά παιχνίδια, αλλά είναι μια λογική έκβαση, ικανοποιητική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ε, υποβάλαμε μια πρόταση στο Συμβούλιο που σας έλεγα για να ληφθεί απόφαση τόσο ώστε να περατωθούν επίσημα ε, οι διαπραγματεύσεις. Αυτό έγινε το 2008. Διευκρινίστηκε πλέον η νομική βάση γιατί θα ξέρετε σίγουρα ότι αναμενόταν και η απόφαση του δικαστηρίου για αυτό το θέμα προς διασαφήνιση της νομικής βάσης. Ε, αυτό έγινε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβει υπόφαση το Συμβούλιο και θα μπορέσει να δώσει συγκατάθεση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σειρά του και χαιρόμαστε που ήδη συζητείται εδώ αυτό το θέμα. Συνεργαζόμαστε στενά με τη ΣΥΠΑ για αυτό το θέμα ε, ούτε είπα, έχουν εφαρμόσει ακόμη το πακέτο ε, αποζημιώσεων Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν βαρύτητα στον τομέα των ε, τυχερών παιχνιδιών. Ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες μελλοντικά στον κλάδο με αυτές τις ε, κινήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, <clears throat> έχει ε, ζητήσει το λόγο πριν ξανακούσουμε τον εισηγητή. Μάλιστα, ένα σύντομο σχόλιο μετά την παρέμβαση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Πράσινη υποστηρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κρίνουμε την είναι λογική ε, προφανώς υπάρχει μια πελώρια βιομηχανία ε, τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στη ΣΥΠΑ και γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικότατα τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτό. Αλλά ας αντλήσουμε και κάποια πολύτιμα διδάγματα. Η Ευρώπη θέλει μέσα στο εμπόριο να ενσωματώσει και άλλες πτυχές ε, πέρα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες αξίες, επιθυμούμε αρχές. τι σημαίνει αυτό λοιπόν ε, στο όργανο ε, επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ και μην ξεχνάτε τους θετικούς και αρνητικούς ε, καταλόγους στην αρχή των διαπραγματεύσεων παραδείγματος χάρη με τον Καναδά. Αν έχουμε αυτή την προσέγγιση των αρνητικών καταλόγων βλέπουμε ήδη ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις που επισύρει μια τέτοια στάση. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, συμφωνώ εν μαζί σας. Ο κύριος Κιούτα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι ανοιχτός προς όλες τις παρατηρήσεις για να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Κατά δεύτερον, όπως ε, προέκυψε και από τις συζητήσεις από τις, ε, με τις μεγαλύτερες ε, εταιρείε του κλάδου, του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, καταλήξαμε σε μία συμφωνία, σε ένα συμπέρασμα, ότι προφανώς αν δεν αποδεχτούμε, αν αναπέμψουμε το ψήφισμα αυτό, ασφαλώς αυτό δεν θα βελτιώσει τα αποτελέσματα των νέων διαπραγματεύσεων. Άρα, εν τέλει, να διευκρινίσω ότι πρόκειται για μια θετική προσέγγιση. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακούσαμε και από τους συναδέλφους, ε, μάλλον ε, συμπεριλάβει τα σχόλια των συναδέλφων, νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα καλό ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούτα, κύριε πρόεδρος. Ε, um, Σας ευχαριστούμε κύριε Κούτας και συγγνώμη για την κολλησιεργία. Δεν υπάρχει προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα δούμε λοιπόν. Το επόμενο θέμα έγιναν κάποιες αλλαγές και τις ανέφερα στην αρχή της συνεδρίασης. Ο κύριος Ντεζίρ θα πρέπει να φύγει και ζήτησε να αλλάξει η σειρά της εξέτασης του θέματος του με τον κύριο Σοντό. Υποθέτω ότι το έχετε συμφωνήσει. Ίσως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ωστόσο γιατί η παρατήρηση αυτή Έφτασε πολύ καθυστερημένα εδώ πέρα στη Γραμματεία και στο Προεδρείο, αλλά να δώσω το λόγο στον κύριο Τεσίρ να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ και τον κύριο Ζαντό για την ε, κατανόησή του. Οι τρει εκθέσει που εξετάσουμε τώρα, Ζαντό, Στενιφιά και η δική μου, ε, συνδέονται μεταξύ του προφανώ, γιατί αφορούν και την ε, συνέπεια τη εμπορική πολιτική δεδομένων των συνολικών στόχων τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση, αλλά και πιο συγκεκριμένα τη λήψη υπόψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων στι εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου και το υπενθυμίζω σε αυτό το σχέδιο έκθεσης βρισκόμαστε απόλυτα στα πλαίσια του πνεύματο των συνθήκων αλλά και του γράμματο, λαμβάνοντα υπόψη του στόχου εμπορική πολιτική. Γιατί υπενθυμίζω ότι το άρθρο 3 τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η εμπορική πολιτική, η κοινή εμπορική πολιτική, θα πρέπει να κυρίω να συμβάλλει στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό μεταξύ των λαών, στο ελεύθερο και ισότιμο εμπόριο, στην κατάρριξη τη φτώχεια, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των παιδιών, καθώ επίση ε, στον αυστηρό σεβασμό ε, του διεθνούς δικαίου και κυρίως ε, των αρχών ε, της Χάρτας των Ηνωμένων, του Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα εμείς και όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι η εμπορική πολιτική σημαίνει κάτι και κάτι άλλο και όχι μόνο ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών όπως άλλωστε είπε και πριν από λίγο ο κύριος Ζαντό και, και θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να μεταφέρει τι προσδοκίε μα για μια παγκοσμιοποίηση που να είναι καλύτερα ρυθμισμένη προ την κατεύθυνση τη αηφόρου ανάπτυξη, τη ανθρώπινη προόδου, του σεβασμού των γενικών αρχών τη διεθνού κοινότητα και ε, του σεβασμού των συμβάσεων των ΗΠΑ ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, προστασία του περιβάλλοντο και ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Η κρίση καταλαβαίνετε ότι ενέτεινε ακόμη περισσότερο την ανάγκη αυτή και η έκθεση ασχολείται με μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή του ζητήματο αυτού, που είναι η σχέση ανάμεσα στην προώθηση τη εταιρική ευθύνη ε, και ε, τη εμπορική πολιτική. Δεν συμπεριλαμβάνει η έκθεση όλε τι προτάσει ε, που, που είχε υποβάλει τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να προβάλλει τι κατευθυντήριε γραμμέ, παράδειγμα, του ΩΣΑ όσον αφορά την εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων για να συμβάλλει στις πρωτοβουλίες καθορισμού ονομασίας των επιχειρήσεων ε, ανάλογα ε, με την εταιρική ευθύνη κτλ. Άλλωστε έχουμε την κυρία Σανιφιέ η οποία έχει τη δική της έκθεση και ο κύριος Αντώ τη δική του που ασχολούνται με τον τρόπο και αυτοί με άλλους τρόπους με τους οποίους στις εμπορικές μας ε, συμφωνίες μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που προτείνουμε και στους εταίρους μας σε θέματα ε, σεβασμού ε, των κανόνων του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασία, προστασία περιβάλλοντο κτλ. Η έκθεση αυτή λοιπόν προτείνει το συνδυασμό δύο τομέων που παρόλο που οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση δεν έχουν συνδυαστεί μέχρι στιγμή. Δηλαδή ε, εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων και βέβαια καταλαβαίνουμε γιατί δεν είχαν συνδυαστεί τα ζητήματα αυτά με την εμπορική πολιτική. Γιατί εδώ μιλάμε για εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων. Ενώ από την άλλη μεριά οι κανόνε του εμπορίου στηρίζονται σε νομικέ δεσμεύσει ε, που αναγνωρίζεται σε διεθνέ επίπεδο. Ε, νομικέ δεσμεύσει των κρατών μελών ε, όπου προβλέπονται και κυρώσει. Η αναστολή, αν θέλετε, των ε, ε, εμπορικών προτιμήσεων σε περίπτωση παραβία των κανόνων αυτών. Στι εταιρικέ ρήτρε, λοιπόν, ή στα κεφάλαια που αναφέρονται στη βιώσιμη ανάπτυξη των εμπορικών συμφωνιών, δεν αναφέρεται η, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, ε, παρά μόνο σε ελάχιστο βαθμό, για παράδειγμα, συμφωνία με την Κορέα και με την Κολομβία και το Περού αλλά ε, εν είδη ε, αναγνώρισης ε, των προϊόντων ισότιμου και δίκαιου εμπορίου. Δεν αναφέρεται λοιπόν σαφώς η στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας της ευθύνη των επιχειρήσεων και όμως νομίζω θα κερδίσουμε αν κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί η βασική εταίρη του σε παγκόσμιο επίπεδο ποιοι είναι. Είναι οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλε πολυεθνικές επιχειρήσει. για τις οποίες η, η, εταιρεία... Η, η κοινωνική ε, ε, ε, ευθύνη των επιχειρήσεων σημαίνει ότι όλα τα, όλοι οι κρίκη των επιχειρήσεων και όχι μόνο οι μητρικέ, αλλά και τα υποκαταστήματα και, και, τα, και οι θηγατρικέ του σε άλλε χώρε, σε, σε χώρε τρίτου κόσμου, εκεί όπου οι κοινωνικοί κανόνε είναι λιγότερο δεσμευτικοί από ό,τι στι ΗΠΑ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζουμε λοιπόν ότι όλα τα σκαλοπάτια μια πολυεθνική επιχείρηση σέβονται αυτού του κανόνε. Ε, ε, φορέ ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτέ οι επιχειρήσει λοιπόν ε, και οι υπεργολάβοι του, οι θηγατρικέ του κτλ. που αποτελούν του βασικού εταίρου και πρωταγωνιστέ του παγκόσμιου εμπορίου, σε αυτέ λοιπόν απευθυνόμαστε και είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα στι εμπορικέ συμφωνίε να αναφέρεται ρητά το πώ θα συνοδεύσουμε τι προσπάθειε τη ανάληψη εταιρική ευθύνη εκ μέρου των επιχειρήσεων. Ε, πώς λοιπόν θα τονίζουμε αυτές που έχουν θετική δράση, έτσι ώστε και οι δύο εταίροι ε, της εμπορικής συμφωνίας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρίτη χώρα ή η ομάδα των τρίτων χωρών, θα φροντίζουμε λοιπόν και οι ΜΕΝ και η ΔΕ, ώστε οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, να τις πείσουμε λοιπόν, εάν δεν έχουν τέτοιες συμπεριφορές, ή ενδεχομένως και να τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Αυτά όσον αφορά τι βασικέ αρχέ ε, τη ε, ε, εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων. Εδώ δεν μιλάμε για έπανα προσδιορισμό του όρου. Έχει οριστεί εδώ και πολλά χρόνια και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία και στον ΟΣΑ εδώ και δέκα χρόνια και στου κόλπου των Ηνωμένων Εθνών. Ε, ξεκινώντας μια πρωτοβουλία του Κόφι Ανάν και στη συνέχεια ε, με το Global Compact, αλλά και εδώ να μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε πολλές ανακοινώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράσινο βιβλίο κτλ. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, υιοθετήσει τις αρχές της εταιρική ευθύνης των επιχειρήσεων. Ποιοι είναι οι άξονες αυτοί. Πρώτα απ' όλα ότι ζητάμε από τις επιχειρήσεις να σέβονται την νομοθεσία. Αυτό είναι προφανές για μας, αλλά εμείς έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο και δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση καταρχήν τουλάχιστον θεωρητικά να μην σέβεται το δίκαιο. Αλλά αυτό αφορά τη συμπεριφορά αυτών των επιχειρήσεων και, των, ε, ε, και της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερος μεγάλος άξονας είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συζητούν με... Ε, ε, τα, τα στοιχεία ε, που υπησέρχονται στι ε, δραστηριότητε του, δηλαδή συνδικάτα αλλά και τοπικές οργανώσεις, για παράδειγμα επιχειρήσει πετρελαϊκέ ή εξόριξης, που είναι πολύ σημαντικό το θέμα της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουν με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους ε, τη συμπεριφορά τους και πώς θα υιοθετήσουν μια συμπεριφορά που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του περιβάλλοντος στο τοπικό επίπεδο ε, των, εργαζομένων έτσι ώστε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της κοινωνίας μας. Υπάρχει λοιπόν ένα τμήμα το οποίο συνδέεται με το νομικό μέρος, νομοθεσία που όλοι θα πρέπει να σέβονται και σήμερα και αυτό αποτελεί ένα μέλημα το οποίο απασχολεί τους πάντες και συμπεριλαμβάνεται στην εργασία για την κοινωνική εταιρική σχέση κατά πολέμηση διαφυγή, ε, διαφθορά κτλ. Και ένα άλλο ε, σημείο το οποίο στηρίζεται σε θελοντική βάση και εδώ μιλάμε για κατά κάποιο τρόπο υπέρβαση τη νομοθεσία. γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για την ίδια την επιχείρηση η ένταξή τη στο ε, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δρά, η ικανότητα τη επιχείρηση να κινητοποιήσει το σύνολο των πρωταγωνιστών την υπηρεσία ε, και άλλων ε, ε, στοιχείων και όχι μόνο για, απο, για αποκόμιση κέρδους. Να καταλάβουν και οι επιχειρήσεις ότι όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση θα ωφελήσουν και τις ίδιες. Τι προτείνουμε λοιπόν. Πρώτον, εκεί όπου ήδη υπάρχει ισχυρή κοινωνική διάσταση σε εμπορικέ συμφωνίε, να συμπεριλάβουμε και την εταιρική ευθύνη. Παράδειγμα, γενικευμένε προτιμήσει συν. Εδώ λοιπόν ήδη υπάρχει το υπόβαθρο για να γίνει κάτι τέτοιο. Προτείνουμε λοιπόν στις, ε, στους εταίρους μας ε, ε, να πέραν δηλαδή αυτών των 25 περίπου διεθνών συμβάσεων που ζητούμε να κυρώσουν, ζητάμε να αναφέρεται συγκεκριμένα να διευκολυνθεί η δικαστική συνεργασία, για παράδειγμα, σε περίπτωση που οι επιχειρήσει δεν σέβονται την νομοθεσία. Δεύτερον, προτείνουμε στην αξιολόγηση αντικτύπου, συχνά το Κοινοβούλιο ζητά αυτές οι αξιολογήσεις αντικτύπου να πραγματοποιούνται με πιο ρεαλιστικό τρόπο εξετάζοντας και τις κοινωνικές επιπτώσεις ε, ε, των εμπορικών συμφωνιών πριν τις διαπραγματεύσεις αλλά και μετά την υλοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας να γίνεται εξέταση ε, του κατά πόσον σέβονται αυτό το ζήτημα οι επιχειρήσεις και σε γενικό επίπεδο, αλλά και συγκεκριμένα τον αντίκτυπο τη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία στι συγκεκριμένε επιχειρήσει στον Α στο Β κλάδο. Αν δούμε δηλαδή ότι μια εμπορική συμφωνία έχει επιπτώσει στην Ελία, εκεί να προσπαθήσουμε να δούμε πώ συγκεκριμένα θα εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσει που δρούν σε συγκεκριμένο τομέα θα σέβονται ε, τι ε, ε, τις νομικέ δεσμεύσει ε, που θα περιλαμβάνει η συμφωνία. Άρα λοιπόν θέλουμε πολύ συγκεκριμένε αξιολογήσει αντικτύπου και να εξετάζεται συγκεκριμένα η επίπτωση συμπεριφορά των επιχειρήσεων και η εξέλιξη τη συμπεριφορά του δυνάμει τη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία και με βάση των αρχών τη κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τρίτη μεγάλη δέσμη προτάσεων στη συμφωνία, στην, πρόταση, στην ε, έκθεση αυτή είναι η συμπερίληψη ρήτρα για κοινωνική ε, εταιρική ευθύνη σε όλε τι μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε και κυρίω τι ε, συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Όσον αφορά αυτέ τι τελευταίε, έχουμε ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη και η φόρο ανάπτυξη. Ε, λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να προσθέσουμε ένα υποκεφάλαιο. Θέλετε μία ρήτρα που να αφορά πιο συγκεκριμένα την ε, κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τι θα συμπεριλαμβάνει η ρήτρα αυτή. Πρώτα απ' όλα αμοιβαία δέσμευση τη Ένωση και των ε, εταίρων για προώθηση τη κοινωνική εταιρική ευθύνη στα πλαίσια τη ε, συμφωνία. Ε, Παρότριση των επιχειρήσεων να αναλάβουν συγκεκριμένε δεσμεύσει με, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνδικάτα, τοπική κοινωνία κτλ. σε θέματα κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τρίτον, δημιουργία σημείων επαφής ακολουθώντα το μοντέλο που εφαρμόστηκε υπό την αιγίδα του ΟΣΑ ε, και εκεί μιλάμε για τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των καταναλωτών κτλ που ε, θα ε, προσφεύγουν ενδεχομένω κατά συμπεριφορών των επιχειρήσεων που έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ή ταυτόχρονα και σημεία όπου θα ενημερώνουν οι επιχειρήσει για το πώ μπορούν να αναπτύξουν τη δράση του προ την κατεύθυνση αυτή. Επίση, δράσει διαφάνεια και υποβολή έκθεση για τι ομάδε και ομίλους, για τι επιχειρήσει και ομίλου επιχειρήσεων. Δηλαδή, υποχρέωση ετήσιου απολογισμού δημόσιου για τι δράσει του συγκεκριμένου τομέα έτσι ώστε να εξετάζεται η συμφωνία ημί με τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν. Γιατί μερικές φορές ε, χρησιμοποιούν οι εταιρείε αυτές τις δεσμεύσεις για λόγους προβολής και μάρκετινγκ. Επίση, ε, υπάρχει κάτι στο οποίο τονίζουν, το οποίο τονίζουν ιδιαίτερα οι συνδικάτε και οργανώσει των πολιτών. Να ε, υπάρξει ε, προληπτική δράση στο συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, να μην μπορούν οι επιχειρήσει να πούν δεν το ήξερα. Δεν ήξερα ότι η δραστηριότητα τη α θηγατρικής μου ή του β υποκαταστήματό μου μπορεί ε, να στηρίζεται σε παιδική εργασία κτλ πρέπει να μπορεί να αποδείξει εκ των προτέρων η επιχείρηση για το ότι παίρνει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε όλοι οι κρίκοι τη αλυσίδα να ε, συμβαδίζουν με τι αρχέ αυτέ. Τέλο, υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει σε περίπτωση παραβίαση, ε, έκδηλη παραβίαση των δεσμεύσεων που έχουν αληφθεί. Ζητάμε πρώτα απ' όλα να υπάρξει μηχανισμός εξέτασης που θα προβλέπεται συμφωνία για περιπτώσεις παραβίασης, να μπορούν να πραγματοποιούνται έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, από εμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το κράτος, εταίρο, αλλά και από ομάδες, ε, ε, ανεξάρτητες ομάδες που θα μπορούσαμε να του αναθέσουμε, όπως για παράδειγμα ε, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας που εξετάζουν τις περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης. Επίσης, ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει επανειλημμένα και εδώ και σε άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Να, ε, παράδειγμα, στην, στην υπόθεση Union Carbide κτλ. Όταν πρόκειται δηλαδή για μεγάλε πολυεθνικέ που δημιουργούν ε, τρομερέ ε, ε βλάβε και που έχουμε ανθρώπινα θύματα κτλ. Ε, ε, και δεν μπορούμε να του βρούμε γιατί δεν βρίσκουν του πραγματικού υπεύθυνου αλλά μόνο του περιεργολάβου. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό ζητάμε να υπάρξουν μηχανισμοί συγκεκριμένη δικαστικής συνεργασίας που να προβλέπονται στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε τη θηγατρική, η οποία είναι για παράδειγμα στην Ευρώπη και να μην μπορεί να ξεφεύγει από τι νομικέ τη υποχρεώσει εάν μία θηγατρική τη παραβίασε την ε, κοινωνική περιοδολογικη νομοθεσία με έκδηλο τρόπο σε, Μια λοιπόν σειρά προτάσει που κάνουμε, δεν θα αναφερθώ σε όλε τι λεπτομέρειε και τελειώνοντα, ε, και εδώ ε, με αυτόν τον τρόπο ε, θέλω να βοηθήσω να περάσουμε και στην επόμενη έκθεση ε, και, και στις λέω ότι πέρα των δικών μας των συμφωνιών, των εμπορικών, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, και στα πολυμερή φόρα να, προ, να, να προωθήσουμε αυτό το συνδυασμό της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης με τις εμπορικές συμφωνίες. Εκεί όπου έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, παράδειγμα στον ΩΣΑ, που είναι φόρουμ ε, προβληματισμού και προώθησης ε, των αρχών της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, στο παγκόσμιο, στην Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας και εμείς, μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε και εμείς εγκρίνει προτάσεις κτλ. να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε λοιπόν ε, και στην ΠΟΕ ε, ένα φόρουμ όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε το συνδυασμό αυτών των αρχών ε, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και στην περίπτωση περιβάλλοντος και εμπορίου οι, επιτροπές, ε, οι αρμόδιες επιτροπές στα πλαίσια της ΠΟΕ έχουν συνεργαστεί με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Ε, ε, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την αξιοπρεπή εργασία ε, θέματα στο οποίο αναφέρεται τώρα και ο ΙΕ, αξιοπρε... αξιοπρεπής εργασία σε όλες τις διαστάσεις και στο όργανο επίλυσης των διαφορών της ΠΟΕ να υπάρξει ε, δυνατότητα υποβολή εκθέσεων από, το Παγκόσμιο Γραφείο, από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία και από άλλα πολυμερή φόρα, αν πρόκειται για το περιβάλλον, για παράδειγμα, για να εξετάζεται ακριβώ η αλληλεπίδραση των εμπορικών κανόνων και τη πιθανή παραβίαση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα για τις παρεμβάσεις σας ε, στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την πρώτη μας συζήτηση, για όλη την εργασία που έγινε μέχρι στιγμής και ελπίζω αυτές οι τρεις εκθέσεις που ελπίζω να ε, ε, εγκριθούν με συνεπή και συμπληρωματικό τρόπο και ελπίζουμε και στις μελλοντικέ μας συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε και αυτές τις προθέσεις να τις μετατρέψουμε σε πραγματικές ρήτρες που θα συμπεριλαμβάνουν τις εμπορικές μας συμφωνίες. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, Χάρλεμ, ε, ο Ντάνιελ. Yeah. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Επειδή ήταν πρόσφατη η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και δυστυχώ δεν μπόρεσε να παρατηθεί εδώ πέρα ο εισηγητής μας. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλέσω όταν αλλάζουμε την ημερήσια διάταξη, όταν πρόκειται για σημαντικό θέμα, να το αναφέρουμε από την προηγούμενη ημέρα, προκειμένου και τα μέλη να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν. Αυτό σε ό,τι αφορά για το μέλλον. Να έχουμε μία μέρα περιθώριο. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο. Διάβασα το Σαββατοκυριακό την έκθεση αυτή και σκέφτηκα τα όσα είχαν συμβεί και βρίσκω πολλά πράγματα στην έκθεση αυτή τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση. Περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, πολλές θετικέ πρωτεβουλίες και θα ήθελα με μεγάλη πλειοψηφία και στην έκθεση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια να υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη, όπου όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και όλο πιο πολλές επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται, θα δυσκολευόμαστε να τις περιορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε πώς ε, οι επιχειρήσεις αυτές θα αντιπεξέρχονται στο ηθικό τους καθήκον, αν θέλετε, σε εθελούσια βάση, αλλά και με κάποιες προδιαγραφές και πώς αυτό θα επηρεάσει και την κατάσταση αν θέλετε, τη ζωή του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και αν οι επιχειρήσεις αυτές τηρήσουν το κοινωνικό τους καθήκον, νομίζω ότι σε πολλούς τομείς, τους οποίους συζητούμε στην παρούσα φάση, δεν θα χρειαστεί να τους ε, συζητήσουμε περαιτέρω, δεν θα χρειαστούμε νομοθετικές προτάσεις οι οποίες συζητιούνται σήμερα, όταν δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις ανταπεξέλθουν και ε, εκπληρώσουν το ηθικό τους καθήκον. Τα σχόλια που έχω να κάνω επικεντρώνονται σε λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση αναφοράς. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση για τις μεγάλες ε, διεθνείς επιχειρήσεις. Κοιτώντα τι γίνεται και με τη συμφωνία με την Νότια Κορέα, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν 10, 15 υπάλληλοι, για παράδειγμα, θα ήθελα να κοιτάξουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα γενικά να συγχαρώ τον εισηγητή και τον ε, εισηγητή Σαΐφη. Νομίζω ότι σε αυτή την ε, νέα περίοδο που ξεκινά θα είμαστε σύμφωνοι για κάποια πολύ βασικά ζητήματα και γενικά είμαι πολύ αισιόδοξο για τις μελλοντικές ε, εργασίες μας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Ντάνιελ, λέει ο πρόεδρος, ο Βίλιαμ. Είναι το μοναδικό φόρουμ που μου ζητείτε να ανάψω το μικρόφωνο μου. Καταρχάς, να πω ότι ο κύριος Σαρίφ είναι πάρα πολύ εύγλωτος και δεν ξέρω αν πέρασε σωστά το μήνυμα. Αλλά να σας πω ότι το εμπόριο είναι εμπόριο. Μιλάμε για εμπορικέ δραστηριότητε, έτσι. Η αρχή που κρύβεται πίσω από το εμπόριο είναι ότι κάποιος ε, κάπου είναι καλύτερο στην παραγωγή ενός προϊόντος από ότι κάποιον άλλο, κάπου αλλού. Αυτό. Δίνει τη δυνατότητα σε εμά τους ανθρώπους να αξιοποιούμε την εξειδίκευσή μας. Και αυτό μας έχει οδηγήσει μετά από αιώνες στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό είναι το εμπόριο, δεν είναι πολιτικό εργαλείο, δεν είναι, ε, θέλετε, καθήκον της πολιτικής να μπλεχτεί σε αυτά. Και δεν θέλω να το θέσω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί σέβομαι πραγματικά τον εισηγητή. Αλλά το πλαίσιο και οι ιδέες που διέπουν τις προτάσεις του κυρίου Ντεζίρ έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ε, περιστάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια και έχουν απορριφθεί επανειλημμένα αυτές οι ιδέες. Και η ιδέα που προτείνει ο κύριος Ντεζίρ είναι σε υπαναχώρηση αν θέλετε. Μιλάμε για μια, ένα, μια απόπειρα να χειραγωγηθεί η εμπορική πολιτική της Ένωσης και μιλάμε για μια τέτοια εμπορική πολιτική την οποία επανελειμμένα έχει απορρίψει το εκλογικό σώμα σε πολλές χώρες και στη δική μας χώρα, στη δική μου χώρα. Τι προτείνετε λοιπόν κύριε Ντεζίρ. Αυτό απομακρύνεται αυτό από αυτό που επιθυμεί το εκλογικό σώμα, ή εκλογής και υπό την έννοια αυτή είναι αντιδημοκρατικό και ξέρω ότι είναι μεγάλος δημοκράτης ο κύριος Ντεζίρη γι' αυτό λοιπόν να το σκεφτεί και από αυτή την άποψη. Στη συνέχεια να διευκρινίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ονομάζουμε πλέον έχει πολλές ε, φιλοδοξίες εδώ και πάρα πολύ καιρό εκτός της επικράτειας της. Και αυτό φαίνεται ότι αποτελεί μία συνέχεια της πολιτικής αυτής για εργαλεία άσκησης ελέγχου εκτός της επικράτειάς της, εκτός των κρατών μελών. Και εγώ ασφαλώς και δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί αυτό ασφαλώς αποτελεί μια αναπηρία για το ευρωπαϊκό εμπόριο. Και μάλιστα μια χρονική στιγμή όπου η οικονομική ισχύ, το εμπόριο κινείται προς Ανατολάς και θα συνεχίσει να κινείται προς Ανατολάς και μάλιστα όλο και πιο γρήγορα αν προτάσεις όπως αυτή εφαρμοστούν και καταστούν νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι πέρα από τον προσωπικό σεβασμό που τρέφω προς τον εισηγητή και τον κύριο Κασπάρη. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική και να τροποποιηθεί σημαντικά η πρόταση αυτή. Να πω ότι σημειώνω αυτό που είπε ο κύριος Ντεζίρ, ότι θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα πεδίο ισότιμων όρων Αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Uh, Ευχαριστώ, Βίλιαμ. Πάντοτε δίνεις έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρειά στη συζήτηση. Ναι, ναι και σαφήνεια. Κριστίν. Δεν πειράζει, συχνά δεν προφέρουν σωστά το όνομά μου. Θα Αφήσω το μικρόφωνο για να μ' ακούν και διερμηνεί, λέει η ομιλήτρια, πέρα από του ε, λοιπού που καταλαβαίνουν τα αγγλικά. I'm very happy ε, καλωσορίζω την έκθεση, χαίρομαι ε, πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η έκθεση. Θα κάνω και κάποιε παρατηρήσει, αλλά ξέρετε η αγγλική μετάφραση μα έφτασε αργά χθε το βράδυ, χθε το απόγευμα, παρότι τη ζητούσα επισταμένα τι τελευταίε μέρε. The other, um, η άλλη συναρμόδια επιτροπή όμως την είχε την έκθεση, οπότε καταλαβαίνετε δύσκολο είναι να γίνει σωστή συζήτηση όταν έχετε στη διάθεση σας το κείμενο εδώ και λίγες ώρες μόνο να πω κάτι και για τον ε, κόμμα του Dartmouth. Είναι ζωτική σημασία να συζητηθεί αυτό το θέμα, διότι πολύ συχνά εταιρείε ε, που δρούν πιο περιορισμένα λόγω των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν διαφορετικά ε, εξ ονόματος της Ένωσης και οι επιπτώσεις, τις επιπτώσεις υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τι έγινε πρόσφατα στην Κολομβία. Είναι Άρα πολύ καλό παράδειγμα παράτυπης συμπεριφοράς ευρωπαϊκών εταιριών σε σχέση με τους εργαζομένους τους που βρίσκονται σε τρίτη χώρα όπου δεν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος για να αναλυφθεί δράση κατά αυτής της συμπεριφοράς ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι δεν μπορεί, εν πάση δεν θέλει να αναλάβει δράση κατά των εταιριών αυτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό μέσα στι συμφωνίε με τι τρίτε χώρε να ενσωματώνουμε και τι ε, κοινωνικέ ρήτρε ε, που θέλουμε να ισχύσουν σε αυτέ τι χώρε ε, όταν δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες ευρωπαϊκές εταιρείες. Εγώ γιατί ανησυχώ. Δεν προβλέπεται εδώ δράση για την υλοποίηση των κανόνων και την εποπτεία, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Ε, βέβαια οφείλουμε να έχουμε επικοδομητική στάση, αλλά πραγματικά πολύ συχνά βλέπουμε υπέροχα πράγματα στις ιστοσελίδες των εταιριών, ε, δηλώσεις ε, που δεν αντιστοιχούν όμως στην πραγματική κατάσταση. Δείτε τι γίνεται στο Δέλτα του Νίγηρα και πώς εμπλέκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, και ποιες είναι οι επιπτώσεις των εμπειρικών δραστηριοτήτων τους επιτόπου. Γι' αυτό σας μιλάω για τον έλεγχο και την εποπτεία και πώς ακριβώς θα καταφέρουμε να ε, επιβάλλουμε μια αξιοπρεπή συμπεριφορά για αυτές τις εταιρείες στις τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε κύριο Σούλτ, Τέιλερ, Λάγγεν και Λίγκφριντ. Αυτοί είναι οι επόμενοι ομιλητές και θα ήθελα να κλείσουμε τον κατάλογο των ε, αγορήτων. Ο κύριο Σούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σύνολο. Οι τρεις εκθέσεις αυτές αποτελούν ένα σύνολο. η περιγραφή της εμπορικής πολιτικής κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και αντίθετα με τον συνάνθρωπο από την Ίσο, θεωρώ ότι είναι πολύ δημοφιλή τα θέματα αυτά, ότι πρόκειται για θέματα τα οποία όντω απασχολούν και τις, ε, το δημόσιο πνεύμα, το ευρύ κοινό. Μιλάει ο κύριος Ντεζίρ για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων η οποία έχει, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε τι γίνεται με τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρετε εκεί πέρα κρύβονται σε πολλές περιπτώσεις η διαφορά και βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, απαιτείται Απαιτούνται συγκεκριμένε ε, ε, διατάξει, ε, απαιτήσει σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευθύνη αυτή. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων σαφών ρυθμίσεων, οι οποίε θα συμπεριληφθούν στην έκθεση. Μία σκέψη επιτρέψτε μου. την οποία θα την εξηγήσω και σε ό,τι αφορά στην έκθεση του κυρίου Ζαντό. Να διευκρινίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η χρονική συγκυρία κατά την οποία συζητούμε τις ε, εκθέσεις αυτές. Μιλήσαμε για την στρατηγική του 2020 και νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι τρεις αυτές εκθέσεις αφορούν την μελλοντική εμπορική πολιτική και συνδέονται με τις προκλήσεις που έχουμε περιγράψει και θα πρέπει να συνδέονται και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι είναι καθήκον και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Άλλη μια σκέψη επιτρέψτε μου κλείνοντας για τις εμπορικές ε, σχέσεις τις οποίες και συζητούμε. Να διευκρινίσουμε ότι όσα αναφέρουμε για το διεθνές εμπόριο αφορούν και το ενδοκινητικό εμπόριο πολλών διεθνών επιχειρήσεων. Γιατί οι διεθνείς επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το ενδοκινητικό τους, ε, τις ενδοκινητικές τους συναλλαγές διέπονται από κάποιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά κοινωνικές ευθύνες και αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών μέσω της καθιέρωσης διαφορετικών προτύπων αναχώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σούλτς, ο κύριος Τέιλορ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η εκδοχή του ε, για, ένα, ε, για, έναν, ε, για ένα τέτοιο πολιτισμό, αναπτυγμένο πολιτισμό του Έλοφ of νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην μειοψηφία. Και κατά την άποψή μου έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον ορισμό και της λέξης αναπτυγμένος αλλά και της λέξης πολιτισμός. νομίζω ότι το όραμά δεν περιλαμβάνει ούτε τη μία ούτε την άλλη λέξη. Ξεκινώ με την έκθεση του κυρίου Ντεζίερ, λοιπόν. Τον ευχαριστώ για την εργασία του. Πραγματικά ε, θα μπορούσε να ε, είχε έρθει λίγο νωρίτερα η αγγλική μετάφραση, ναι. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα ήμουν ιδιαίτερα ε, ευγνώμων. Αν στο, στο μέλλον δεν έχουμε ε, τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, στην έκθεση περιλαμβάνονται διάφοροι τομεί ε, διάφορα σημεία τα οποία ε, ε, τονίζουν το γεγονό ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη θα πρέπει να συνδέεται με τι εμπορικέ συμφωνίε. Οι εμπορικέ συμφωνίε πρέπει να έχουν και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το γεγονό ότι η εθελοντική προσέγγιση, ο εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας έχουν μέχρι στιγμή αποτύχει και δεν έχουν καταλήξει σε σημαντικέ αλλαγέ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η κοινωνική εταιρική ευθύνη. Και η συνεργασία ε, θα πρέπει να, η εμπορική συνεργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και λογοδοσία μέσω τη δικαστική οδού, αν προκύπτει. Ε, μπορεί να γίνει εργασία ε, και βεβαίω όλοι θα υποβάλουμε τροπολογίε, αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε το χρόνο να καταλάβουμε τι ακριβώ περιλαμβάνει η έκθεση λεπτομερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπέρτ. Ευχαριστώ και εγώ καλωσορίζω την έκθεση. Ρητά, συνάδελφοι, γιατί θεωρώ ότι αν θέλουμε να πάρουμε σε σοβαρά τη συνθήκη της Λισαβόνας, τις αξίες οι οποίες εμπεριέχονται και προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της συνθήκης της Λισαβόνας, δεν μπορούμε να διαιρέσουμε στα δύο την πολιτική μας για τις επιχειρήσεις και να πούμε ότι α, το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο δεν μας αφορά καθόλου γιατί δεν είναι ε, δεν εντάσσεται στο ιστορικό της Ένωσης γιατί μιλάμε για ένα σύνολο αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν καλώς ορίζω την καθιέρωση σαφών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτές. Και αυτό θα πρέπει να μπει ως ρήτρα πραγματικά σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες αυτές. Αυτό που με απασχολεί είναι ο έλεγχος της στήρισης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτών και πώς θα μπορούσε να συμμετάχει πιο έντονα η κοινωνία των πολιτών. Στο 12 ή και F αναφέρεται ο έλεγχος και υποχρέωση αναφοράς στην κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ορίζονται και κάποιες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Τα συνδικάτα, ίσως οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να ορίζονται οι ομάδες αυτές προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν κατά πόσο τηρούνται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ανομαλίες να μπορούν να τις επισημάνουν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάχιτφριντ. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Νομίζω ότι η έκθεση του συναδέλφου Ντεζίρ είναι πραγματικά εξαιρετική. Επί του περιεχομένου ε, περιλαμβάνει όλα όσα εκπροσωπώ. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω τα οποία ακούσαμε. Εννοείται ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί πολιτική και όχι μόνο εμπόριο. Κοιτώντας την ε, συνολική ιστορία του ανθρώπου βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν πολιτικοί σκοποί πίσω από κάθε δράση και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Ευρωπαϊκή θέλει, Ένωση θέλει να ασκήσει εμπορική πολιτική όχι για να εκμεταλλευτεί άλλους όπως πολύ συχνά έχει γίνει στην ιστορία αλλά για να ταχθεί υπέρ των ανθρώπινων αξιών θα πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Και όταν μιλάμε για δημοκρατική νομιμότητα, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι κάθε κρατος μέλος εθελούσια, εθελοντικά επέλεξε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναγκάστηκε, δεν εξαναγκάστηκε καμία χώρα Άρα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίζονται τα θέματα. Δεν ξέρω πώς ήρθε εδώ πέρα στην ε, επιτροπή μας ο συνάδελφο Δάτμα στο κοινοβούλιο μας. Εγώ πάντως είμαι δημοκρατικά εκλεγμένος και αυτό σκοπεύω να κάνω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν πρόκειται να επισέλθουμε στο δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο εκλέγονται ε, οι ερωτήσει σήμερα. Κοιτάξτε, συνήθω όταν κλείνω ένα κατάλογο μιλητών, τον κλείνω έτσι. Αλλά επειδή δεν έχει συνηθίσει να είμαι εγώ πρόεδρο, σου δίνω 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση αρχής και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ντεσίρ ε, για την ε, συνεισφορά του, για το σχέδιο έκθεσης. Βλέπω ότι επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Σαΐφη. Βρίσκονται πάρα πολύ κοντά αυτές οι δύο εκθέσεις. Και θα έλεγα ότι ο μείζον όρος, η μείζον διατύπωση είναι αυτή που αναφέρεται στην, ε, στον τίτλο της έκθεσης κυρίας Σαΐφη. Και θα έλεγα ότι η έκθεση του κυρίου Ντεσίρ θα όφιλε να τελεί σε σχέση υπαλληλία ε, έναντι της εκθέσεως της κυρίας Σαΐφη. Δηλαδή θα έβλεπα ε, κανονικά να έχουμε ένα κείμενο. Αυτή η πολυδιάσπαση ε, δεν ξέρω γιατί πρέπει να γίνεται. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Μου θυμίζει λίγο με όλο το σεβασμό που έχω στην Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων, στην Επιτροπή ΦΑΜ, μου θυμίζει λίγο εκθέσεις εκείνης της Επιτροπής. Και τελειώνοντας, θέλω να πω Βεβαίω πρέπει να υπάρχουν ρήτρε, αλλά πρόκειται για ρήτρε οι οποίε περιβάλλονται έναν διακηρυκτικό χαρακτήρα, έχουν declaratory character και από τη στιγμή που δεν έχουν τα στοιχεία, τα ποιοτικά του κανόνα δικαίου, ίσω κουβεντιάζουμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τη... σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Um, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, να σας δώσω το λόγο και σας δώσω συγγνώμη την πρώτη φορά δεν είπα σωστά το όνομά σας. Σα ευχαριστώ. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση του κύριου Τεσίρ και μας δίνει πολύ υλικό για σκέψη. Ε, ήρθε επίσης στην κατάλληλη χρονική στιγμή, ιδιαίτερα διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για, τις, για τη μελλοντική επενδυτική πολιτική και υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση βεβαίως στο σημείο αυτό. Μιλάμε για πολυεθνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό. Επίσης έρχεται τη χρονική στιγμή όπου ε, πολλές γενικές διευθύνσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, εργάζονται για μια νέα ανακοίνωση πάνω στην κοινωνική εταιρική ευθύνη και μην ξεχνάμε ότι ε, αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη του ΩΣΑ εργάζονται για επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΩΣΑ. Και βεβαίως θα ληφθεί υπόψη. και αυτό το ζήτημα της αλυσίδας εφοδιασμού. Άρα λοιπόν έχουμε ε, πολλά χρήσιμα στοιχεία για να τα σκεφτούμε και αυτή τη στιγμή τα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Βεβαίω είναι πολύ δύσκολο ο τομέα αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τη σωστή ισορροπία αυτή τη στιγμή ε, η προσέγγιση μας είναι κυρίως εθελοντική. Και βεβαίως αυτό μπορεί να είναι ε, πιο αποτελεσματικό σε ορισμένε περιπτώσει έναντι άλλων. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσει σέβονται απόλυτα τον νόμο και έχουν μια σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά, αλλά ταυτόχρονα να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να ε, αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ε, και να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτούς άξονες. Ταυτόχρονα πρέπει να εξετάσουμε ε, και τα πρακτικά στοιχεία. Εδώ μιλάμε για, νομική, για μια νομική σύμβαση ανάμεσα σε δύο κράτη όταν μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες και για πολυεθνικές που, που δεν είναι πάντα μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αλλά μπορεί να είναι και μικρές εταιρείες ε, όπως για παράδειγμα ε, ξένοι επενδυτές. Είναι πολύ πολύπλοκα τα ζητήματα αυτά και στην έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχονται πολλά χρήσιμα στοιχεία τα οποία εμεί θα λάβουμε υπόψη με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ευχαριστώ. Χάρλεμ, μπορεί να συνοψίσει πολύ γρήγορα. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Ναι, ευχαριστώ, Ρομπέρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σα λόγια και για τι προτάσει σα αυτέ για να συμπληρώσουμε και να διευκρινίσουμε περαιτέρω τα στοιχεία τη έκθεση. Ευχαριστώ τον κύριο Κάσπαρη για την υποστήριξή του. Πραγματικά πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να διακρίνουμε αυτό το οποίο ζητάμε από τι πολύ μεγάλε επιχειρήσει και αυτό το οποίο αφορά τι ε, μικρού μεγέθου επιχειρήσει, που όμω και αυτέ έχουν δράσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και μικρομεσαίε επιχειρήσει που δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο και που βεβαίω δεν έχουν τη διαμέσα με τι μεγάλε πολυεθνικέ για να υπόκεινται στι ίδιε υποχρεώσει. Βεβαίω πρέπει να σέβονται τι δεσμεύσει και του κανόνε, αλλά ίσω εδώ, για παράδειγμα, σε επίπεδο ε, αυτή τη έκθεση που ζητάμε δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Ε, τώρα, κοιτάξτε, ε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε συζητήσει και στην καφετέρια. Αλλά βεβαίω το εμπόριο είναι εμπόριο. Και όταν λέτε στην ουσία αυτό το οποίο μετράει είναι να λάβουμε υπόψη αυτός που, αυτός ε, που μπορεί να παράγει κάτι άλλο με καλύτερο τρόπο αλλού. Ναι, μπορεί βεβαίω κανείς να παράγει πιο αποδοτικά ε, χρησιμοποιώντας παιδιά, ε, φυλακισμένους, να καταστρέφει το περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα ούτε για μας αλλά ούτε για τις χώρες εταίρους. Άρα μην ξεχνάμε και το ίδιο το πνεύμα της συνθήκης. Το θύμισε και ο κύριος Λάγκε. Το πρώτο άρθρο, εγώ παρέφησα το άρθρο 3 πριν από λίγο η εμπορική πολιτική πράγματι θα πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο γενικότερο ε, τη εξωτερική μα πολιτική. Πρέπει να αποτελεί έναν τρόπο για προώθηση τη εμπορική δραστηριότητα ε, κτλ. Αλλά και άλλων κανόνων ε, στι συναλλαγέ μα για ένα καλύτερο κόσμο. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι ε, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίε ε, των πολιτών. Ε, οι εκλογέ κερδίζονται, χάνονται, είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι σαφέ, ότι η κοινή γνώμη και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι το, το γεγονό αυτό. Δηλαδή ότι οι εμπορικέ συμφωνίε δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο για το συμφέρον των επιχειρήσεων και ει βάρο των κοινωνιών, αλλά να προωθούν τι αξίε μα και τι αρχέ μα. Αυτό προσδοκούν όλοι οι πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπέρντερ έχει δίκιο όταν μιλάει για το θέμα του ελέγχου και για τον τρόπο με τον οποίο όλε αυτέ οι δεσμεύσει που αναλαμβάνονται από τι επιχειρήσει υλοποιούνται συγκεκριμένα. Και για το πώ εμεί επαληθεύουμε τη συμβατότητα ανάμεσα στι δεσμεύσει και στην πρακτική. Ναι, αυτό είναι κεντρικού κεντρική σημασία θέμα στην, στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. Και εδώ θα πρέπει κάπω να, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο όσον αφορά τι προτάσει. Ο κ. Σούλτ μίλησε για τη σχέση με τη στρατηγική 2020 και με την παγκόσμια στρατηγική, αν θέλετε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δίκιο. Και τόνισε επίση και το, ε, το ζήτημα του ελέγχου και τη αποτελεσματικότητα ε, των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. Ο κύριος Τέιλορ απάντησε τον κύριο Ντάρτμουθ και είπε ότι οι πορισμένε ε, πτυχέ. Ναι, ναι, μάλλον είναι αλήθεια ε, ότι υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά το καθαρά εθελοντικό επίπεδο και το δεσμευτικό. Ναι, το είπα και εγώ. Η πρώτη διάσταση είναι να ζητάμε από τι επιχειρήσει να σέβονται την νομοθεσία. Αλλά η νομοθεσία δεν ε, είναι προαιρετική και το είπε ο κ. Κασπάρη πριν από λίγο αν όλα πήγαιναν καλά και, όλοι, ε, και όλα δούλευαν ρολόι και όλοι σέβονταν σε εθελοντική βάση τι υποχρεώσει του, ε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά αν δεν υπάρχουν κανόνες, ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν γίνονται πάντα σωστά σε εθελοντική βάση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και δεσμευτική διάσταση και διάσταση υποχρέωση. Και ίσω πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτή τη στιγμή. Η, η εμπλοκή της εταιρείας των πολιτών και, ε, ε είναι βασικό για, για, για λόγους ελέγχου. Αυτό το θέμα της, των σημείων επαφής ε, λειτουργεί καλά ε, αλλού, περισσότερο, αλλού καλύτερα, αλλού χειρότερα. Το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία όπου ε, οι πολίτες μπορούν να, να φέρουν αυτά τα οποία διαπιστώνουν είναι πολύ σημαντικό γιατί προσδίδουμε αξιοπιστία στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. Βεβαίω συμφωνώ στην απάντηση που έδωσε ο κύριο Ντάρτμουθ για την πολιτική διάσταση εμπορική πολιτική και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή τη. Βεβαίω, Γι' αυτό συνδέεται και με τι άλλε εκθέσει, όχι μόνο του κ. Ζαντό, αλλά με την άλλη έκθεση που επίση προετοιμάζει για τι επενδύσει. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη νέα διάσταση της ε, πολιτικής των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμπόριο με την αυστηρή έννοια του όρου, επενδύσεις, αλλά και σύνδεση με τις εργασίες που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική εταιρική ευθύνη στους κόλπους του ΟΣΑ αλλά και ε, των Ηνωμένων Εθνών, όπου περιμένουμε και μια νέα έκθεση η οποία θα αφορά κυρίως το ζήτημα των αλυσίδων εφοδιασμού Δηλαδή να ξεπερνά την ε, αυστηρή δομή τη ε, μητρική επιχείρηση, αλλά να καλύπτει όλε τι αλυσίδε εφοδιασμού. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι σχετικά σύντομη, αλλά θα μα επιτρέψει να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την εργασία αυτή. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. you, Ευχαριστούμε, κύριε Ντεζίρ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν είναι 5 Οκτωβρίου, είστε σίγουρος. Εμένα είχα την εντύπωση ότι η προθεσμία έχει οριστεί για την 5η Οκτωβρίου. Πρόεδρος, το πρόβλημα είναι η μετάφραση. Μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο αν το επιθυμείτε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε πρόβλημα με τη μετάφραση ο κύριος Ντεζίρ. Νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Υπάρχει και μεταξύ των δύο και συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι συνάδελφοι, αλλά χρειάζεται χρόνος όχι μόνο για τη μετάφραση, αλλά και για τη σύνταξη των, τροπολογιών. Ε, ε, θα συμφωνήσω. Ε, πήρα χτες το βράδυ ε, την έκθεση στα αγγλικά και τι θα έχουμε δύο μέρες μόνο για να εμπεδώσουμε το περιεχόμενό της. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Ωραία, 5η Οκτωβρίου τότε. Συμφωνείτε όλοι. Ε, ναι, δεν διαφωνώ, αλλά αποκλείεται να τα προλάβουμε όλα μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου. Ε, Πολλοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την έκθεση, κυρίως λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο συναδελφός μας ο κύριος Ντεσίν Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να οριστεί η προθεσμία στην 5η ε, Οκτωβρίου. Ντάνιελ. Νομίζω ότι το νωρίτερο που μπορούμε να επιβάλλουμε είναι η 5η οτι το νωρίτερα αλλά να θέσω και το εξή θέμα στις αρχές του έτους μοιράσαμε στις ομάδες τις εκθέσεις και αφήσαμε χρόνο προκειμένου να προετοιμάσουν και οι συγκητές καλές εκθέσεις. Το θέμα είναι το εξής. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να περάσει στην Ολομέλη το Νοέμβριο το θέμα αυτό. Ή μήπως θα μπορούσαμε να αφήσουμε και λίγο πιο πολύ χρόνο. Ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν νέες ε, εκθέσει πρωτοβουλία, αλλά αν θα μπορούσαμε να περιμενουμε τρει τρει-τέσσερι εβδομάδε, δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε, ε, δεν θα αποτελούσε πρόβλημα αυτό. Και κοιτώντας και την διάταξη της Ολομέλειας, ε, νομίζω ότι υπάρχει χρόνος. Άρα, να βάλουμε την 5η Οκτωβρίου ή να δώσουμε πιο πολύ χρόνο. Ναι, συμφωνήσαμε, Πρόεδρε λέει ο πρόεδρο Ντάνιελ για την 5η Οκτωβρίου. Το πρόβλημα είναι η 25η Οκτωβρίου, όχι η Ολομέλεια. Δεν ξέρω Συμφωνείτε να ορίσουμε λοιπόν την 5η Οκτωβρίου ως προθεσμία. Oui, euh, merci, euh, cher... Ευχαριστώ Ρομπέρ, αγαπητέ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αγλέμ Ντεζίρ για ε, την σκληρή εργασία του για την έκθεση αυτή και θα συμφωνήσω μαζί του. Οι τρεις εκθέσεις, η δική του, η έκθεση του κυρίου Ζαντό και η δική μου ε, είναι αλληλένδετες. Συμφωνώ με την απάντηση που έδωσε προς τον ε, κύριο Ντάρτμουντ. Ε, ναι, το εμπόριο είναι εμπόριο, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Θα ήθελα τώρα να περάσω στα ουσιαστικά σημεία της έκθεσης. Ε, όπως σας έχω ήδη πει, έχουμε διτή προσέγγιση με στην έκθεση. Πρώτον, μέσα στις διεθνείς συμφωνίες ε, θέλουμε να ενσωματώσουμε και να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμόζονται οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες με καλύτερο τρόπο. Επίσης, αμοιβαιότητα των ε, ανταλλαγών πρέπει να κατοχυρωθεί με τους διάφορους εμπορικούς μας εταίρους. Και από αυτή την πλευρά ευθυγραμμιζόμαστε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16 ε, Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών συμφώνησαν ότι είναι καθοριστική σημασία να αναπτύξουμε την εμπορική συνεργασία με στρατηγικού εταίρου για να δώσουμε νέα τόνο στην οικονομία, να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Είπαν επίση ότι είναι απαραίτητο η εμπορική αυτή πολιτική να χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα. Μέσα στο σχέδιο δεν ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα παντού, ούτε στι φτωχέ χώρε μπορούμε να επιβάλλουμε του ίδιου κανόνε όπω και στι πλούσιε χώρε. Ε, πονούμε κάποιε προτάσει όμω για να αποφύγουμε καταστάσει αθέμητου εμπορίου. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε τρεις επιλώνες, η τήρηση, η πολυμερή στήριση των κανόνων, διμερή στήριση των κανόνων και μονομερή στήριση τους. Ε, για το πολυμερές επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες αδρές γραμμές ε, για την πολυμερή συνεργασία και συγκεκριμένες προτάσεις ε, για την συνεργασία στα κοινωνικά ζητήματα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας Φερρυπίν που θα αποφαίνεται κάθε φορά που διαπιστώνεται παραβίαση ή τίθεται κάποιο ζήτημα βασικών κανόνων χρόνων κοινωνικών. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες ε, πρασίνων τεχνολογιών να ε, συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το άρθρο 31 ε, της δήλωσης της Δόχα και τέλος προτείνεται να δημιουργήσουμε έναν διεθνή οργανισμό περιβάλλοντος χάρη στον οποίο θα υπάρξει τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων. Το περιβαλλοντικό δίκαιο και το εργατικό δίκαιο θα πρέπει να έχουν ισότιμη θέση όπως και το εμπορικό δίκαιο. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ή και ένας μελλοντικός περιβαλλοντικός παγκόσμιος οργανισμός θα μπορούσαν να παρέμβουν γιατί όχι και στις εμπορικές διαφορές μέσω προδικαστικών ερωτημάτων. Ε, σε διμέρες τώρα επίπεδο, το σχέδιό μας ε, συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση πιο συγκεκριμένα ε, το ε, αντικτύπου επί της βιώσιμης ανάπτυξης όλων αυτών των μέτρων. Θεωρούμε ότι με το που θα αρχίσει να ισχύει η συμφωνία μπορεί να γίνει η αξιολόγηση. Το σχέδιο προτείνει κυρίως στο πλαίσιο των Συμφωνίων Ελευθέρων Συναλλαγών να εφαρμόζουμε το, το, την αρχή της ευελιξίας και της σταδιακής αντιμετώπισης κατά την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Ένα ζήτημα δηλαδή απαλής πίεση που στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών θα κατοχυρώνει την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων. Στο σημείο 15 όμως η έκθεση μιλάει για τους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων ε, και μιλάει για την διαιτησία, για τα φόρα ανταλλαγών και διαπραγματεύσεων της κοινωνίας των πολιτών και προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής κατά των συμφωνιών με δυνατότητα επιβολής προστήμων εάν δεν υπάρχει τήρηση του κεφαλαίου περιβιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Οπότε θα ζητήσω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί γιατί διαπραγματεύεται τώρα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τον Καναδά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα, καλό θα είναι να συζητηθεί το θέμα των ακυρώσεων ε, για την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και του Διεθνούς, ε, Εργατικού Δικαίου. Τέλος σε μονομερές επίπεδο στη διαδικασία αναθεώρησης ε, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσάρμοσε τα κριτήρια για να μπορεί κάποιο να υποφεληθεί από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων του ώστε λιγότερο ανεπτυγμένε και προηγμένε χώρε να μπορέσουν να υποφεληθούν και να υπάρχουν μηχανισμοί αντιπαράθεση σύγκριση, ε, διαφανεί μηχανισμοί για τη χορήγηση των προτιμήσεων δυνάμει αυτού του συστήματο. Ιδού λοιπόν σχολίασα όλα τα ουσιαστικά ζητήματα και μέσα στην ε, έκθεσή μου ε, θέλησα να, περά, να ξεφύγω από ένα απλό ευχολόγιο. Είναι δύσκολο το ζήτημα και είναι σημαντικό σε τούτου να έχουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στο εμπόριο. δηλαδή πώ θέλει ε, η Ευρώπη να προχωρήσει στα πλαίσια τη στρατηγική 2020. Ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στο εμπόριο και στις υπόλοιπες δράσεις ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση, Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επικρατήσει συνοχή ανάμεσα στι τρει εκθέσει του κ. Ντεζίου, του κ. Ζαντό και τη δική και να, είμαστε, να δώσουμε αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία και να περάσουμε ένα ενιαίο μήνυμα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Ρόμπερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τόκια για το σχέδιο έκθεσής της όπου τονίζει τις ε, βασικές ανησυχίες ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Ε, η Τόκια, όπως σωστά είπε, ότι είναι αλληλένδετες οι εκθέσεις αυτές, οι τρεις εκθέσεις, η δική της, η έκθεση του Γιάννη και η έκθεση του Χάρλεμ. Βλέπουμε τις βασικές προτεραιότητες που συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοι Δηλαδή θέλουμε να είναι δίκαιη η ανάπτυξη, επωφελής για όλους, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου, ενώ ε, τονώνουμε το εμπόριο. Πέραν αυτών των γενικών παρατηρήσεων, δεν έχω πολλά ειδικά σχόλια. Ε, θα έχω άλλη μία γενική παρατήρηση και θα επανέλθω και το απόγευμα στην ακρόαση. Το Global Europe, ε, η παγκόσμια Ευρώπη δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών μας τελικά. Ε, και η στρατηγική 2020 και η νέα εμπορική πολιτική δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών μας σε αυτό το τομέα, διότι παραμένει αναλύωτη η φιλοσοφία, δηλαδή άνοιγμα των αγορών θεωρείται αυτό αυτοσκοπός, ο μοναδικός αυτοσκοπός και χαίρομαι από τις δηλώσεις ε, του Επιτρόπου στην αντίστοιχη ε, ακρόαση που έγινε δεν μπορεί να επαρκέσει από μόνο του το εμπόριο. Συγχαίρω την Τόκια Safe, λοιπόν για την έκθεσή της. Ε, σίγουρα θα την ξανασυζητήσουμε. Ε, θα επιμείνω για ένα σημείο. Αυτό το θέμα των ε, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι νομικώς ε, δεσμευτικά αυτά τα πρότυπα. Αλλιώ ε, δεν ε, αξίζει να κάνουμε υπέροχες εξαγγελίες επί σειρά ετών χωρίς να είμαστε σε θέση όμως να επιβάλλουμε την εφαρμογή τους. Πρέπει να είναι νομικώς δεσμευτικά αυτά τα πρότυπα. Αυτό είναι ο πυρήνας του ζητήματος και κάτι άλλο. Ε, δεν θα πρέπει να δώσουμε αυτή την προστατευτική εικόνα χρησιμοποιώντας ε, τέτοια ε, ένδικα μέσα. Δεν πρόκειται για κυρώσεις, πρόκειται για δημιουργία ουσιαστικής εταιρικής σχέσης και πλαισίου πραγματικού διαλόγου. Οφείλουμε να έχουμε θετική προσέγγιση και πάνω απ' όλα θα πρόσθετα εγώ ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειε μα. Θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε και να προσθέσω επίση ότι η Τόκια μέσα στην έκθεσή τη αναφέρει σε κάτι που εντάξει δεν μου δημιουργεί ανησυχίε απαραίτητα, αλλά μου δημιουργεί ερωτηματικά. Αυτή η αρχή τη αμοιβαιότητα. αναφέρεται στην αμοιβαιότητα έχοντα ένα ευρύτατο όραμα που καλύπτει όλες τις τρίτες ε, χώρε. Νομίζω ότι υπάρχει μια συμμετρία μέσα στην έκθεση λοιπόν. Θα πρέπει να προσέξουμε αναχώρηση χώρα δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες σχέσεις με όλες τις τρίτες χώρες. Ε, αυτά είναι ήδη προκατακτικών σχολείων ε, για την έκθεση της ε, Τόκια. Σε συγχαίρω. Πραγματικά είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ, Κέντα. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές, Τάιλερ, Ζαντό και Μπέρλερ και κλείνω τον κατάλογο. Παρακαλώ. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω κοιόδης ε, για τους ε, ε, πράσινους για αυτή την έκθεση θέλω να συγχαρώ την εισηγητρία για την εξαιρετική της εργασία. Η έκθεση αυτή δεν μπορούσε να έρθει μια πλέον κατάλληλη στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε προ το σχεδίασή τη νέα εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ζητήματα όπω κοινωνική εταιρική ευθύνη, ε, περιβαλλοντικά πρότυπα ε, να ε, διαπνέουν απόλυτα τη νέα εμπορική πολιτική. Χαίρομαι γιατί αναφέρεστε σε, σε δεσμευτικά κεφάλαια για την αηφόρο ανάπτυξη. Εξαιρετική επίση η ιδέα τη αιρεσιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών με τη πρόσβαση στην αγορά να εξαρτάται από τι επιδόσει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Χαίρομαι ε, με αυτή την υπόδειξη για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού για το περιβάλλον. Επίσης, ε, το σχέδιο έκθεσης προτείνει ε, ενίσχυση ε, του καθεστώτος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, Εκεί όπου θα μπορούσαν να αλλάξουν ορισμένα σημεία ε, στην έκθεση, να σα πω το εξή. Δεν συμφωνώ απόλυτα με την συγκίτρια για το ότι οι ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στη συμφωνία με την Κολομβία αρκούν. Αυτή ε, η τυπική διατύπωση που δεν σημαίνει τίποτα θα πρέπει να μετατραπεί σε δεσμευτική, σε δεσμευτική υποχρέωση με κυρώσεις. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ε, τη Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου για το εμπόριο και το περιβάλλον θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά. Και σύμφωνα με τον συνάδελφο και εισηγητή ε, για την έκθεση ε, ε, για την αλλαγή του κλίματος, τον κύριο Γιαντό, προτείνουμε να αλλάξει μέρος της διατύπωσης παραγράφου 9 όσον αφορά τα εργαλεία για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης θα ήθελα να υπάρξει όθηση για ένα διεθνές νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό σε πολυμερές επίπεδο και σε διμερές επίπεδο νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για επεξεργασία ε, των κριτηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στα πλαίσια ε, του νέου νομικού πλαισίου για τις δεσμεύσεις ως μέρος των νέων υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει σαφής λογοδοσία και κυρώσεις για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επίσης, η ανάγκη εξέτασης ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, ε, των κρατικών προμηθειών, υπηρεσιών κτλ. για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ελλείψεις ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίδραση στο κλίμα. Και τέλος πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος όσον αφορά το θέμα της πρόσβασης των θυμάτων στα δικαστηρία, της προστασίας των θυμάτων και της άμεσης αποκατάστασής τους θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Απλά και μόνο θέλω να πω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή που γίνεται σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών για τι επιπτώσει τη παγκοσμιοποίηση, για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν ορισμένοι συμπολίτε μα όσον αφορά την καλύτερη κατανόησή του ε, για την εμπορική πολιτική, το κοινωνικό ντάμπινγκ, το περιβαλλοντολογικό ντάμπινγκ, το νομισματικό ή φορολογικό ντάμπινγκ κτλ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αφορά άμεσα ε, τι εργασίε τη Επιτροπή μα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά την ομάδα των Πρασίνων, εμεί πιστεύουμε ότι η, η, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πράγματι, ε, όπω είπε ε, ε, και ο Καντεραδίφη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα της αμοιβαιότητας ε, που αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, ε, στην αιτιολογική σκέψη Βρισκόμαστε σε επίπεδο ε, αμοιβαιότητας δικαίου ή αμοιβαιότητας εμπορικών ε, πλεονεκτημάτων, αμοιβαιότητας δικαιωμάτων ή εμπορικών πλεονεκτημάτων. Ε, τι, πού βρίσκεται η συμμετρία και ε, τι επίπεδο αμοιβαιότητας έχουμε πραγματικά. Επίσης και εμείς είπαμε στην κυρία Σαϊφή ε, τις απόψεις μας και θέλουμε να αλλάξει η παράγραφος 9. Προφανώς θέλουμε να αναφέρεται σαφώς ότι οι, ε, διαπραγματεύσει για το κλίμα θα πρέπει να γίνουν πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ΟΗΕ και όχι στα πλαίσια αυτά τα οποία θα μπορούσε ε, να δημιουργηθεί εντύπωση ότι αναφέρεται μέσα από το κείμενο, δηλαδή ότι σε, σε επίπεδο G20 για το κλίμα. Ευχαριστώ. Κάθριν. Εκτός μικροφώνου. αυτή η συζήτηση συνδέεται με την ε, προηγούμενη και είναι ε, ιδιαίτερα επίκαιρη, αλλά δημιουργεί κάποια σύγχυση. Γιατί ορισμένα από τα ζητήματα ε, συμπεριλαμβάνονται και στι δύο εκθέσει. Πάντω, όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση, κατά την άποψή μου, εδώ περιέχονται τα βασικά ε, θέματα που είναι τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Απόλυτα ζωτική σημασία, λοιπόν, όχι μόνο για καλέ εμπορικέ πρακτικέ, αλλά και για την ίδια την επιβίωση και τη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη, τη, τη ζωή των ανθρώπων στον πλανήτη αν θέλετε. Πολύ συχνά Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στι δύο διαστάσει, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Όταν μιλάμε για του αυτόχτονε ε, και για την καταστροφή του δάσου, μιλάμε και για ανθρώπινε ζωέ και για περιβάλλον. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τι δύο έννοιε. Και ε, χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που, αλλά για άλλη μια φορά ερχόμαστε στο θέμα της ε, υλοποίησης, εφαρμογής, της συμμόρφωσης, ε, της παρακολούθησης ε, και της εργασίας σε προδιαπραγματευτικό επίπεδο. Εκεί πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα. Κυρίως θα μιλάμε για περιβαλλοντικά πρότυπα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε σε μια τρίτη χώρα δεν θέλουμε να καταστρέψει τα δάση σου. Γιατί μπορεί ε, το δάσο ε, να αποτελεί και η ξυλία να αποτελεί το μοναδικό του πόρο, αν θέλετε, και αντικείμενο εμπορία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και λογικοί, αλλά και να φροντίζουμε και το θέμα τη συμμόρφωση. Αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για πόρου των αναπτυσσόμενων χωρών και είπα, ε, ε, ακολουθούν μια διαδικασία εξέτασης ε, του, του αντιτίμου για αυτά τα αγαθά. Ε, ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ να είστε σύντομος γιατί αργήσατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Καταλαβαίνω ότι δείχνετε κατανόηση όμως. Δεν με ικανοποιεί η έκθεση αυτή την κορυφή του παγόβουνου πετυχαίνει σε ό,τι αφορά τους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά πρότυπα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά να θεωρώ ότι μπαίνει στον πυρήνα των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του εμπορίου. Θεωρώ ότι τα συμφέροντα, τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτά τα οποία υπογραμμίζονται στο κείμενο αυτό και όχι τόσο το θέμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Η επικρατεί μεγάλη ασάφεια σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, δεν προτείνει ουσιαστικές διαφορές, αλλαγές. Θεωρώ ότι η πραγματικότητα του ευρωπαϊκού εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών ανησυχιών καταδεικνύονται από τις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συνήθισαν με την Κολομβία και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αποδεχτεί σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή και τη σύναψη συμφωνίας με μια χώρα όπου παραβιάζονται κατάφορα τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τη σύναψη συμφωνιών θα πρέπει να προαπαιτούμε τουλάχιστον να ευθυρούνται ε, η απέτηση η, τα συμβαλώμενα μέρη να έχουν ε, υπογράψει τις συνθήκες του, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Και επίσης να υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζόμενων και τέλος, Πρόεδρε, επέστρεψα πρόσφατα από μία αντιπροσωπεία στο Καζακστάν, όπου δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, αλλά που πολλές ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και βγάζουν μεγάλο κέρδος σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα. Και βλέπουμε ποια είναι η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων που είναι κατάφοροι. Αυτό φυσικά δυστυχώ δεν απέτρεψε τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το να προβαίνουν σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι είναι μεγάλο το κενό μεταξύ του ιδεατού και της πραγματικότητας. Και αυτό θα πρέπει να τονίσουμε. Ευχαριστώ, Τζο. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε την ευκαιρία για να κάνω και εγώ κάποια σχόλια για την έκθεση της κυρίας Σέιφη. Θα είναι σύντομα τα σχόλιά μου. Θα προσπαθήσω βέβαια να απαντήσω στις ερωτήσεις που απίθυνε στην Επιτροπή κυρία Σέιφη, κυρίως για τις κυρώσεις. Η έκθεση της κυρίας Σέφη είναι σχετικά πλήρης αλλά και σύντομη και περιεκτική. Υπάρχουν στοιχεία μέσα στην έκθεση που από τη δικιά μας ε, τη σκοπιά επιβεβαιώνουν απλώς στοιχεία που ήδη έχουν υλοποιηθεί. Αντίθετα υπάρχουν ε, και άλλα στοιχεία που προτείνουν ενίσχυση του συστήματος, ε, βελτίωση της δράσης των εφισταμένων εργαλείων. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ιδέες για μελλοντικέ δράσεις και πρωτοβουλίες. Πράγματα που σήμερα δηλαδή δεν έχουν ήδη γίνει από τα θεσμικά όργανα. Φυσικά δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τους νέους προσανατολισμούς, τις νέες ιδέες, τις προτάσεις που γίνονται για το μέλλον. Τούτου λεξέντως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια τεχνικά και πρακτικά ζητήματα που όμως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, κυρίως για τα πρόστιμα. Η κυρία Σέφη ε, μας ζήτησε να κάνουμε ένα σχόλιο για την ε, βορειοαμερικανική πρακτική. Τρία μοντέλα υπάρχουν, τέσσερα για να είμαι πιο ακριβής, αλλά εγώ θα σχολιάσω τα τρία. Σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να ενσηματώσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα στις συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών. Το πρώτο μοντέλο προβλέπει νομικές υποχρεώσεις που συνοδεύονται από διαδικασία των παρακολούθησης, ελέγχου, ε, με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ε, αυτό ε, προάγουμε εμείς από πλευράς Επιτροπής. Υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο τώρα, όπου οι νομικές υποχρεώσεις συνοδεύονται από την υποχρέωση, την δυνατότητα ανάκλησης των παραχωρήσεων, δηλαδή αν υπάρχει παραβίαση των δειγμάτων εργαζομένων για να κερδίσει μια χώρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να μπορούμε εμείς να δράσουμε με τα εμπορικά εργαλεία αμερικανικό μοντέλο. Τώρα τρίτον, καναδικό, καναδέζικο μοντέλο για, τις, ε, τα εργατικά πρότυπα, δηλαδή εμπορικές προτιμήσεις με επιβολή οικονομικών ε, κυρώσεων που θα απαιτούνται ε, από την νομολογία των τρίτων χωρών που παραβιάζουν της ε, διατάξεις του μοντέλου. Αυτές είναι οι τρεις εναλλακτικέ λύσεις, αλλά όπως σας έλεγα ε, υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά πρακτικά και τεχνικά ζητήματα λόγω των οποίων ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Καναδοί τελικά χρησιμοποίησαν ε, το σύστημα επιβολής κυρώσεων ή αντιπίνων διότι ε, δεν είχαν αρκετά εργαλεία στη διάθεσή τους ε, ούτως ώστε να υποχρεώσουν ε, τις τρίτες χώρες να βρούνε και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να καταβάλουν τα πρόστιμα ή δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν να αναπτυχθεί η νομολογία και το ένομο σύστημα αυτών των τρίτων χωρών για να ενσωματώσει αυτές τις νέες ρήτρες. Τέλος να μην μακρηγορώ αλλά κατά τη γνώμη μας θα έλεγα συνοψίζοντας πως η συζήτησή μας ε, θα πρέπει να καλύψει όλες τις τεχνικές και πολιτικές πτυχές ε, τα πρακτικά ζητήματα επίσης ούτως ώστε να ε, συνειδητοποιήσουμε τελικά προς ποιο μοντέλο προσανατολιζόμαστε. Για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σημαστική συμπερίληψη της σχετικής ρήτρας μέσα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες θα λέγαμε ότι υπό την, ε, τον τίτλο Εμπορική Συμφωνία προβλέπονται πολλά διαφορετικά ε, πράγματα. Δηλαδή, ε, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα έχουμε μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Μπορεί να χαρακτηριστεί και εμπορική αυτή η συμφωνία. Νομίζουμε πάντως δεν είναι απολύτως απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε αυτόματα μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί έχουμε και τις συμφωνίε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, εμπεριέχουν, αν θέλετε, τις εμπορικές ε, συμφωνίε, Οπότε δεν χρειάζεται επικάλυψη, εφόσον προβλέπεται ήδη αυτή η ρήτρα. Ήθελα, θέλησα να το διευκρινίσω αυτό και να προτείνω ίσως ότι η συστηματική συμπερίληψη αυτής της ρήτρας τελικά δεν θα πρέπει να θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση απαραίτητα. Ευχαριστούμε. Αυτά ήθελα να πω. Πρόεδρος, ε, θα ακούσουμε την Τόκια Σαϊφή, την εισηγήτριά μας και πάλι για να κλείσει η συζήτηση. Ναι, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει από ό,τι βλέπω. Να ε, καθησυχάσω το Γιάννη Ξαντό. Όλες οι κλιματικές διαπραγματεύσεις σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθούν και όχι στο G20. Κύριε Τέλερ, Είπατε ότι έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Ορίστε, μόλις ακούσατε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκω την ισορροπία μέσα στην έκθεσή μου. Υπάρχουν ε, θέματα ε, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλησα να φορτώσω την έκθεση. Ε, Καντέρα Ρίφ, μα στο σημείο 13 και 15 μιλούμε για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων, αλλά μιλάει για υποχρεωτικό μηχανισμού μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων. Θέλω να διευκρινίσω τι ακριβώς εννοείται. Θα μπορούσαμε εξάλλου να ζητήσουμε και μία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κύριε Αρίφε, τι εννοείτε μιλώντας για δεσμευτικά δικαιοδοτικά όργανα, γιατί εγώ στο σημείο 13 και 15 το αναπτύσσω το θέμα. Απάντηση. Ίσως να αναφερθούμε και στις ε, ε, Ευχαριστώ Τόκια που ε, μίλησε συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα και έτσι Πρόεδρε μπορώ και εγώ να σα πω ότι όπω και για την προηγούμενη έκθεση θα πρέπει να αναβάλουμε μέχρι την 5η Οκτωβρίου την ε, προθεσμία υποβολή τροπολογιών και στι 13 Οκτωβρίου έχουμε και ένα συνέδριο για το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία για διοργάνωση του σεμιναρίου και σα προσκαλώ. Ε, συγγνώμη, κάνατε μία ερώτηση, ε, κυρία Σέιφη. Ναι, ναι, όχι, ήθελα να ευχαριστήσω απλώς τους συναδέλφους ε, πριν κλείσω για τη συνεργασία τους. Ευχαριστούμε, κυρία Σέιφη. Η προθεσμία, λοιπόν, είναι η 5η Οκτωβρίου για την υποβολή των ε, τροπολογιών στις 6 το απόγευμα και για τις δύο εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Άλλη μία λοιπόν διεθνής εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, Γιάννικ Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν αρχίσω θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον ε, πρόσωπο της Επιτροπής για τις απαντήσεις που μας έδωσε. Ήταν ιδιαίτερα πολιτικής φύσεως θα έλεγα όσον αφορά τη συζήτηση αυτή και αυτό νομίζω ότι είναι καλό. Είναι καλό, σε τελευταία ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθά ε, για να οικοδομήσουμε τη συζήτησή μα Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν μ' δεν πειράζει. Τέλειωσε το θέμα, άρα δεν ενδιαφέρεται. Τέλο πάντων, δεν είναι σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα του εμπορίου και των κλιματικών αλλαγών, ήδη κάναμε δύο συζητήσει επί του θέματος και είχαμε τη μετάφραση την περασμένη εβδομάδα. Απλά και μόνο να πω και να αναφέρω ορισμένα σημεία τα οποία τα βρίσκουμε και στην ίδια την έκθεση. Νομίζω ότι ορισμένα ε, αιτήματα και ερωτήματα που έγιναν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι σημαντικά και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ, ε, τις Επιτροπές ΔΕΒΕ και ΕΝΒΗ, για τη συμβολή τους στη συζήτηση της έκθεσης. Προφανώς λοιπόν εδώ, όπως αναφέρθηκε ήδη, κυρίως στην έκθεση της κυρίας Σαϊφή, εδώ πρέπει να δούμε πόσο σημαντική είναι η σύνδεση ε, ε, των γραμματιών των ε, συμφωνιών αυτών των διεθνών με την εργασία της ΕΠΟΕ. θα τα βρείτε όλα αυτά μέσα στο, στην έκθεση. Πιο συγκεκριμένα, ενίσχυση της ανάμεσα στο εμπόριο και στην προστασία του κλίματος. Προφανώς θέλουμε να υπάρξει ε, αύξηση των συναλλαγών όσον αφορά τα αγαθά και τι υπηρεσίε περιβαλλοντολογική φύσεω που βοηθούν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό τόσο επί της τεχνολογίας όσο και επί των ε, προϊόντων και των υπηρεσιών περιβαλλοντολογική φύσεως να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία επιτρέπουν να ορίσουμε τι είναι τελικά το ένα αγαθό ή μια υπηρεσία περιβαντολογικής φύσεως. Και όλα αυτά σα λέω στα πλαίσια καταπολέμηση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή και της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά τη μεταφορά της τεχνολογίας. Όλοι γνωρίζουμε, παρόλο που δεν έχουμε σήμερα ε, μαζικά ε, τεχνολογικά μέσα που να βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Απ' την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι αν εντείνουμε όπως αποτελεί απέτηση των επιστημόνων ε, τον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής θα υπάρξουν πολύ περισσότερε συναλλαγέ ε, και ανταλλαγέ τεχνολογίας. Αλλά εδώ ε, πρέπει να προσέξουμε μην βρεθούμε σε κάποια περιορισμένα πλαίσια ε, όπου χώρες θα βρεθούν εκτός. Διότι η τεχνολογία είτε καλύπτει από δίπλωμα βρεστεχνία, είτε είναι περιορισμένη χρήση και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες χώρες, κυρίως ανεψόμενε χώρε. Το θέμα των ε, επιδοτήσεων ε, για ε, την, ε, την ενέργεια. Εδώ έχουμε υποδείξει στις 20 και άλλων. Ξέρουμε όλοι σήμερα ότι όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα βρισκόμαστε γύρω στα 500-600 δις δολάρια όσον αφορά την επιδότηση στον τομέα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για απόλυτη συμβατότητα με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα θέλαμε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αναλάβει την ηγεσία. Και άλλωστε αυτή θα γίνει και μια συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το θέμα ε, της ε, διαφυγής άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο ανακύπτει διαρκώς. Μόλις ε, συζητάμε τις φιλοδοξίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. έχουμε ε, ε, το, το, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παίρνουμε το 20 ε, και θέλουμε εδώ να υπάρξουν συγκεκριμένα μέσα για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκοί κλάδοι που θα αποτελέσουν που θα, είναι αντικείμενο απειλή εάν η, Ευρω... η Ευρώπη γίνει περισσότερο φιλόδοξη. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να φύγουμε από αυτά τα φαντάσματα ε, που συνδέονται ε, με τη διαφυγή άνθρακα. Δεν μιλάμε για 164 ε, κλάδους που απειλούνται, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και αξιόπιστοι. Να σταματήσουμε λοιπόν αυτή τη λογική ε, του ΓΙΣΕ που σημαίνει ότι δεχόμαστε όλους τους οικονομικούς ε, ε, κλάδους που ζητούν παρέκκληση. Κυρίως από το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων ένταξη σε διεθνέ επίπεδο και κυρίω σε επίπεδο ΠΟΕ ε, αυτή τη διαφοροποίηση των προϊόντων ανάλογα με, την, ε, ε, με τις κλιματικές τους, τις στο κλίμα. Αυτό βεβαίω συνδέεται με συγκεκριμένου κανόνε, dumping κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα αυτό σε επίπεδο ΠΟΕ και βεβαίω παρόλο που οι, οι σε επίπεδο ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντικέ εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη, κυρίως ε, με αυτά τα οποία έγιναν για τα ευρωκαύσιμα, δεν μπορεί να εντάσσει στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες κριτήρια βιωσιμότητας. Αντίθετα, σας θυμίζω μάλιστα ότι αν δεν κάνω λάθος, οι Ηνωμένε Πολιτείε μόλις ενσωμάτωσαν στις εμπορικές του σχέσεις με το Κογκό ένα δελτίο ταυτότητας, αν θέλετε, όλων των ε, ε, των πολιτήμων μετάλλων που εισάγονται στη ΣΥΠΑ, έτσι ώστε να εξφαλθεί το γεγονό ότι δεν χρηματοδοτείται με τον τρόπο αυτό, ε, δεν χρηματοδοτούνται οι πόλεμοι στην περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ΥΠΑ μπορούν να το κάνουν. Μα και εμεί μπορούμε. Και μπορούμε από σήμερα να συμπεριλάβουμε στοιχεία τα οποία αφορούν τι διαδικασίε και μεθόδου παραγωγή. Πάντα όσον αφορά τι εμπορικέ συμφωνίε που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν, ε, αμφισβη, δεν τίθεται σε κίνδυνο ο αγώνας κατά πολέμηση κλιματικής αλλαγής, ότι δεν υποβασμίζονται οι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν την καταπολέμηση της ε, ε, κλιματικής αλλαγής. Εδώ μιλάμε για την αποψήλωση των δασών, για τη γεωργία, για τα μοντέλα τα οποία άμεσα ή έμεσα υποστηρίζουμε, κυρίως στις χώρες του Νότου. Και τελειώνω, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο, γιατί βλέπω ότι ανυπομονείτε. Βεβαίω. Καταλαβαίνω. Ε, ε, το, δεν, καταλαβαίνω ε, ότι είστε συγκεκριμένα καθήκοντας πρόεδρος. Δεν αφήνω το, το, το ενδιαφέρον σας για το θέμα μου, αλίμονο. Πάντω, όταν για παράδειγμα διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά, δεν αμφισβητούμε τον κατά κάποιο τρόπο δογματικό τρόπο με τον οποίο, ε, ε, τον ακολουθεί αυτός αυτή η χώρα. Έχουμε για παράδειγμα το Ontario Green Act ε, που ε, θέτει συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά σε τοπικό επίπεδο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα το σημείο αυτό. Επίση, επίσης, ε, οι ε, μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μα θα πρέπει, και τελειώνω εδώ, να συμπεριλαμβάνουμε σε εμπορικές ε, συμφωνίε να έχουμε ένα κεφάλαιο για το κλίμα έτσι ώστε να αξιολογείται το ισοζύγιο άνθρακα. Και αν είναι πολύ κακέ οι επιδόσει όσον αφορά το ισοζύγιο του άνθρακα, ε, να προσαρμόζεται κατά συνέπεια και κατά ακολουθία και η εμπορική συμφωνία. Γίνονται και άλλε συζητήσει ε, σε άλλε επιτροπέ για, το, για, για, για καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότηση. Και εδώ βεβαίω ε, το θέμα αφορά άμεσα το ζήτημα κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ, για το χρόνο που μου έδωσε για να σα παρουσιάσω την έκθεση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γιάννη. Τρει ομιλητέ έχω. Λίκφριντ, Κασπάρη και Κλάτφελ. Και Τζο Χίγκιν. Κοιτάξτε, αυτή τη φορά κλείνω τον κατάλογο, έτσι. Προσπαθώ να είμαι σύντομο γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μιλάω εξ μου. αντικαθιστώ τον ε, κύριο Κιούτες. Αλλά ασφαλώ και συμφωνώ με όλα όσα λέει, με όλα όσα εκφράζει. Να πω λοιπόν τα εξή. Υπήρξαν κάποιες βασικές στιγμές ε, κατά τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να μιλήσει με μία φωνή στην Κοπεχάγη το 2009 για παράδειγμα. Αν αυτού, αντί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, διαδραμάτισε ένα ρόλο ο οποίο τελικά δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να δραματίσει πιο σημαντικό ρόλο η Ένωση στην καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος και σε όλες τις σχετικές πολιτικές, γιατί υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών και της Στρατηγική της Ευρώπης για την αλλαγή του κλίματο. Οι εκπομπέ σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ και το διεθνέ εμπόριο επηρεάζουν ασφαλώς έχουν γίνει θετικά βήματα για την ε, κοινωνία σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, το οποίο φυσικά είναι υποφελέ για την κοινωνία, αλλά συνεπάγεται και περιβαλλοντικέ ε, επιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε τι ευθύνε μα από το διεθνέ εμπόριο σε ό,τι αφορά τι τις ε, χώρε, τι αναπτυσσόμενε και τι χώρε τις βιομηχανοποιημένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον ΠΟΕ και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισάγει στις εμπορικές ε, συμφωνίες κάποιες ρήτρε δεσμευτικέ σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε επίπεδο ΠΟΕ και το GAP, GAP Plus θα πρέπει να λάβει υπόψη τέτοια περιβαλλοντικά πρότυπα. Και τέλος θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες διεθνείς συμφωνίες για την περιβαλλοντική διάσταση και εγώ και ο κύριος Κιούτας είμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας υπηρεσίας παγκόσμιας για το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να πω ότι Προς τη σωστή κατεύθυνση οδεύει η έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα επειδή η αρχική έκθεση για το θέμα αυτό, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ήταν αρκετά αρνητική. Κινούταν προς την κατεύθυνση του ότι το εμπόριο είναι αρνητικό για το περιβάλλον. Θεωρώ ότι τώρα είναι πιο ισορροπημένη η έκθεση. Τονίζονται και οι θετικές πτυχές. Μιλάμε και για περιβαλλοντικά προϊόντα, για τα σύγχρονα προϊόντα της τεχνολογίας, τα οποία μας ε, βοηθούν να μειώνουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι θετικά βήματα αυτά. Ένα θέμα πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τον Οκτώβριο σε ό,τι αφορά των διασυνοριακών αντισταθμίσεων. Το έχουμε συζητήσει αυτό και το, αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην έκθεση ΣΑΕΦΗ, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια τέτοια λύση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορικοί μας εταίροι δεν θα κάνουν περιβαλλοντικό, κλιματικό dumping. Θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση ανάλογη με την διατύπωση της συναδέλφου ΣΑΕΦΗ στο σημείο 9 όπως για παράδειγμα και σε μια διατύπωση τύπου της διατύπωσης που έχει επιλέξει ο κ. Ζαντό. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε σχετική συμφωνία. Κατά τα άλλα, να σας ευχαριστήσω γιατί θεωρώ ότι είναι καλή η έκθεση και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον να γίνουν πολλές αλλαγές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλο και πιο πολύ Ακούμε διάφορα σχόλια σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του, της εμπορικής πολιτικής και ότι το εμπόριο του μέλλοντος θα βασίζεται πιο πολύ στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και όχι στην φθηνή εργασία. Προς το παρόν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να να αποφύγουν τη φορολογία ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις για την αξιοποίηση της ενέργειας. Ιδιαίτερα βλέπουμε ότι υπάρχουν περικοπές στην τιμή της, ε, του ρεύματο και επίσης επιδοτείται το κόστος των καυσίμων όταν το καύσιμο αυτό προορίζεται για εξαγωγή. Την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καινούργια εμπορική της πολιτική σχεδιάζει να απορριθμίσει, να απελευθερώσει την εισαγωγή προϊόντων μεταλλουργίας τα οποία είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας. Προφανώς αυτό οδηγεί σε κατάσταση προς την Απανατολή και θα υπάρχουν πολλές πιο πολλές εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή ε, των ίδιων προϊόντων στο τμήμα αυτό, στο μέρος αυτό του κόσμου. Αυτό φυσικά δεν βοηθάει τον αγώνα μας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, γιατί τα σχέδια αυτά με την κατάσταση ουσιαστικά συμβάλλουν στην αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και μιλάμε για τα κράτη εκείνα τα οποία αποτρέπουν και παρεμποδίζουν, παρακολύουν τις ε, πρωτοβουλίες της Κοπενχάγης. Αυτά τα κράτη είναι τα κράτη που τελικά έχουν πλέον εκτίματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και όχι τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ε, μιλητής, ο συναδελφός Χέλμον Σούλτς, παρακολουθεί το θέμα αυτό και θα ήθελε να πει ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί με την έκθεση του κυρίου Ζαντό ότι η καινούργια στρατηγική για το εμπόριο του 2020 θα πρέπει να λαμβάνει τα στοιχεία της έκθεσης αυτής υπόψη και τα βασικά ευρήματα. Και τέλος, εξ μου, Πρόεδρε, να πω ότι το θέμα της συνέπειας, της συνοχής, το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή. Μιλάμε για συνοχή μεταξύ την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, των αξιών της που έχει δηλώσει σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ε, θέλουμε συνοχή μεταξύ της πραγματικότητας του εμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος αφετέρου. Ωστόσο, το εμπόριο που διεξάγεται από τις μεγάλες οντότητες ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες ε, επιχειρήσεις δεν επιδεικνύει καμία συνέπεια. Πώς γίνεται να έχουμε μεταφορές φρούτων για παράδειγμα από μία μακρινή χώρα και να υπάρχουν αεροπλάνα εμπορευμάτων που να κάνουν πολλαπλέ διαδρομέ κάθε μέρα. Σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ για να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείτε τι μεταφορέ γίνονται σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα απορροκυπευτικά. Μιλάμε για μαζικό κέρδο, το οποίο ντρέπουν οι μεγάλε εταιρείε με χαοτικό τρόπο και δυστυχώ ε, θα συνεχίσει να πλήττει το περιβάλλον αυτή η πρακτική. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ Τζο και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Διαβάσαμε την έκθεση και παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο και επικοδομητικό το έγγραφό σας. Ε, τροφοδοτείται η συζήτηση με τις συστάσεις και τις απόψεις που εκφράζονται μέσα στην έκθεση. Ε, κοιτάξτε, έχουμε και εμείς παρεμφερείς απόψεις, αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ε, σημεία όπου διαφοροποιούμεθα λίγο από πλευράς Επιτροπής. Τρία-τέσσερα στοιχεία θα αναφέρω για να κάνω κάποια σύντομα σχόλια ε, για την διαρροή άνθρακα. Θεωρούμε ότι η κατάσταση απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση διότι σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις. Ε, θυμηθείτε και την ανακοίνωση που εκδώσαμε το Μάιο για αυτό το θέμα και υπάρχουν διατάξεις για την διαρροή άνθρακα που, θα αρχίσουν, που άρχισαν να ισχύουν από το 2009 άρα επαρκούν προς το παρόν αλλά θα γίνουν και άλλες αξιολογήσεις στο μεταξύ. Τα PPM, η μεθόδη παραγωγής, ε, διαφοροποίηση ως προς την παραγωγή παραγωγή είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα ανάμεσα στα μέλη του ΠΟΕ γιατί υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ε, οπότε η προοπτική για να καταλήξουμε σε συμφωνία ή το ενδεχόμενο ε, ε, ίδια ερμηνεία ή παρέκκληση από τους κανόνες είναι ιδιαίτερα ίσχνες και έχουμε και τις διμερείς συμφωνίες που πρέπει να καλύπτουν αυτά τα κριτήρια και θυμηθείτε ότι υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων για τα βιοκαύσιμα τώρα ε, έχουμε μεγάλες προκλήσεις και εμείς ε, και είπα σε, όπως προς τις εμπορικές συναλλαγές. Ε, για τις ρήτρες τώρα, τις κλιματικές σχετικά με τις τοπικές ρήτρες και τη συμπερίληψή τους σε συμφωνίες, θα έλεγα το ίδιο όπως και για τα αντίστοιχα μέτρα, δηλαδή θα δημιουργηθεί επικοινωνία κίνδυνο προηγούμενο αν επιτρέψουμε να ε, ε, καταρτιστούν και να εφαρμοστούν ε, τέτοιες πολιτικές. Σχετικά με τη χρηματοδότηση των μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές είναι σημαντικό να επικρατήσει η διαφάνεια ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι οικονομικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Εμείς θα ε, παρουσιάσουμε στην Κανκούν μια εμπεριστατωμένη έκθεση και επίσης θέλουμε να συλλέξουμε σχετικές πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Θα θέλατε σύντομα να σχολιάσετε αυτή την παρέμβαση. θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή τους θεωρώ ότι το θετικό είναι ότι μας, έχουμε δύο επιλογές ουσιαστικά ε, δοθεί τη κατάστασεις ή θα παραμείνουν ε, στο ίδιο ύψος οι προσδοκίες ε, που έχουμε για τις κλιματικές αλλαγές ή θα ε, τις τροποποιήσουμε αλλά αν τις τροποποιήσουμε θα χρειαστούν και τα εργαλεία ούτως ώστε αν χρειαστεί να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τις απειλούμενες ε, βιομηχανίες. Ε, τώρα για τη δεύτερη εναλλακτική λύση, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών όπως ε, αναφέρει ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο Ε, καταλαβαίνω τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έκθεση ε, της Επιτροπής, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια δόση κριτικής σε σχέση με αυτά που έγιναν για την οδηγία ΕΤΕΣ σχετικά με την διαρροή άνθρακα και Θα έλεγα ότι ο στόχος είναι ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογή ε, των ε, αποκλήσεων και των ε, δωρεάν ποσοστώσεων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κοινή διεθνή δέσμευση. Όπως είπε και ο κύριος Χάσπαρη και όπως γράφει και η κυρία Σαϊφή στην έκθεσή της, το πλεονέκτημα για τη μέθοδο του άνθρακα είναι ότι βοηθάει τις ε, χώρες εταίρους ε, να είναι ε, πιο φιλόδοξες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή και ενδιαφέρουσα ιδέα. Ευχαριστώ Γιάννη και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι μαντέψτε η 5η Οκτωβρίου όπως και για τις υπόλοιπες εκθέσεις και έχετε την αμέριστη υποστήριξή μου όπως ξέρετε. Πολύ ωραία. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μαύρη Θάλασσα. Ε, κύριος Καζάκα, ευχαριστώ Ροπέρ. Ε, βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο ε, στην ε, διάθεσή μας, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Κάναμε ήδη μία πρώτη ανταλλαγή, μία ακρόαση πιο συγκεκριμένα που διοργάνωσε ο συνάδελφος από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την ίδια τη στρατηγική, για την ίδια την έκθεση, στα πλαίσια της οποίας μου εδόθη η ευκαιρία να τοποθετηθώ για την στρατηγική αυτή. Θα ήθελα όμως ε, σε αδρές γραμμές να σας παρουσιάσω τις προτάσεις κλειδιά ε, που εισηγούμε εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ε, θα είναι το περιεχόμενο της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για αυτό το θέμα. Πρώτον, Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οι εμπλακόμενες χώρες επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό. Είναι λίγοι ανευαίσθητες χώρες και υπήρξαν ολέθριες επιπτώσεις ως προς τα αναπτυξιακά ποσοστά που μέχρι τότε ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 6%. Θα πρότεινα λοιπόν να ενισχυθεί η εταιρική σχέση κυρίως στα πλαίσια ε, του, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του εξήνου Πόντου για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ολέθριες επιπτώσεις ενισχύοντας λοιπόν τις χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές ρυθμίσεις για να αυξηθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια ως προς τον προϋπολογισμό. Δεύτερον, ε, η συνέργεια του εξήνου Πόντου που δρομολογήθηκε το 2007 έδωσε νέα όθηση στην περιφερειακή συνεργασία ε, πλην όμως Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, για να αποφύγουμε επικάλυψη παρεμφερών περιφερειακών πρωτοβουλειών στον τομέα αυτό. Η συνέργεια του Ευξήνου Πόντου σε σχέση με την ανατολική εταιρική σχέση, παραδείγματο χάρη. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να γνωρίζουμε ε, ποιε είναι οι προτεραιότητε τη εκάστοτε πρωτοβουλία, ούτω ώστε να αποκομίζουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Εξήνου Ποντού είναι μία, έχει έναν απολογισμό 20 ετή θετικό ε, το 2012 είναι η 20η επέτειος και θα είναι η καλή ευκαιρία για να κάνουμε ένα νέο απολογισμό και να προτείνουμε ενδεχομένως κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις για να βελτιστοποιήσουμε τη δομή και τη λειτουργία του οργανισμού ε, για κάποια όργανα όπως η Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Συμβούλιο των Επιχειρήσεων. Τέταρτον, η συνέργεια της, ε, του ευξήνου πόντου, ε, κατά τη γνώμη μου, έχει θετικό αντίκτυπο ε, ως προς τις στοχευμένες προτεραιότητες της, δηλαδή μεταφορές ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι πρωτοβουλίες και να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να προαγάγουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οικοδόμηση στρατηγικών υποδομών όπως ο, το δικό δίκτυο γύρω από τον Εύξηνο Πόντο καθώς και τις θαλάσσιες οδούς μεριμνώντας όμως ώστε να μην θέσουμε εν κινδύνο την ε, ασφάλεια, τη θαλάσσια ασφάλεια. Ε, τέλος, Συνάδελφοι, όλο ένα και περισσότερε χώρε συμμετέχουν σε αυτόν τον Περιφερειακό Οργανισμό Οικονομική Συνεργασία ε, πλην δύο χωρών και δείχνει αυτό ευθυγράμμιση ω προ τους οικονομικούς κανόνες του οργανισμού αυτού και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Προτείνω λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση προ όλε τι χώρε τη περιοχή αυτή να συνεχίσουν τι προσπάθειέ και να άρουν όλου του εμπορικού φραγμού ή καταδεικνύοντας και μία αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Κόζα. Τρεις ομιλητές και έκλεισε ο κατάλογος. Ο Τζούμουλς, ευχαριστώ, πρόεδρε. Ξεκινώ λέγοντάς ότι πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η καταδεικνύοντας και μια αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Κοζά. Τρεις ομιλητές και έκλεισε ο κατάλογος. Ο Τζούλς, ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ξεκινώ λέγοντάς ότι πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση αυτή που ακούσαμε και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο για το ότι και η ακρόαση που έγινε πριν από δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ καλή η ακρόαση. Στην ουσία λοιπόν πιστεύω ότι έδωσε πολύ καλά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της ιδέας της μετατόπισης από τη συνέργεια σε στρατηγική στο τομέα της, ε, του ευξήνου πόντου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ε, ε, ε αλλά είναι αλλά έχει και συγκεκριμένη παρουσία, έτσι, ε, από το 2007 ε, στον εύξηνο πόντο. Τώρα, ορισμένε υποδείξει όσον αφορά την επικάλυψη και το φόβο ότι ορισμένε πρωτοβουλίε θα μπορούσαν ε, να αποτελούν αντικείμενο επικάλυψη είναι βάσιμη φόβη αυτή. Πάντα όμω εγώ είμαι υπέρ ε, των θετικών εκφράσεων. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε για συμπληρωματικότητα. Μελλοντική στρατηγική λοιπόν για τον εύξηνο πόντο που θα πρέπει να συμπληρώνει τι άλλε πρωτοβουλίε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, πρωτοβουλίε για τη Μεσόγειο, ε, τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία κτλ. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, οικονομική στήριξη, εδώ πιστεύω ότι η στρατηγική, η μελλοντική στρατηγική για τον εύχρονο πόντο θα πρέπει να, συμπε, ε, να συμπεριλαμβάνει και τη χρηματοδοτική στήριξη, από τα διάφορα μέσα, από το πρωτεξιακό μέσο, ε, έτσι ώστε να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν συγκεκριμένε ε, χρηματοδοτικέ και οικονομικέ προοπτικέ για το μέλλον. Και τέλο, μία παρατήρηση, μάλλον μία πρόταση για την ενέργεια. Επειδή είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ενέργειας για την περιοχή, νομίζω ότι η ολόκληρη περιοχή θα πρέπει να στοχεύει στην ε, ε, ολοκλήρωση στη νέα ευρωπαϊκή ε, αγορά ενέργειας, όπως, όπως, όπως και αν την ονομάσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για μερικά ή ορισμένα συγκεκριμένα σχέδια, το Ναμπούκο, το South Stream, το σχέδιο για το υγροποιημένο αέριο κτλ. Για το LPG. Ενδεικτικά τα αναφέρω. Θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε και εκεί ονομαστικά και ίσως να μιλήσουμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Γιατί εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο οι υδρογονάθρακες αλλά και αυτά ε, τα ανανεώσιμα ε, προϊόντα, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι πολύ σημαντικέ για την αηφόρο ανάπτυξη αλλά και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Πράγμα εξίσου σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζούλ. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση πολύ σωστά τονίζει το θέμα της ανάπτυξης των υποδομών και θα ήθελα να ε, ξεκαθαρίζει ε, ακόμα περισσότερο ε, την, την σημασία που έχει η ανάπτυξη των λιμένων στην περιοχή. Επίχει και αναφέρω συγκεκριμένα την Κωνσταντζα στη Ρουμανία μην ξεχνάτε ε, τη στρατηγική σημασία του, ε, ε, τη στρατηγική θέση του συγκεκριμένου λιμανιού. Όταν έχουμε μεταφορά αγαθών από την Ανατολή προς τη Δύση, παρόλο που το λιμάνι της Κωνσταντζας ενδείκνεται ιδιαίτερα, δεν το χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιούνται άλλα λιμάνια στη Δυτική Ευρώπη. Για να φτάσουν τα αγαθά στη Βουδαπέστη ή στο Βουκουρέστη ε, κάνουν όλο το, ε, το, γύρο της Ευρώπης Και δεν χρησιμοποιούμε το λιμάνι αυτό. Ακριβώς γιατί οι εγκαταστάσεις είναι απαρχιωμένε. Απαιτείται δεκαπλάσιο χρόνος για να φορτωθεί ένα ε, πλοίο συγκεκριμένο λιμάνι σε σχέση με το λιμάνι του Ρότερνταμ. Και μην ξεχνάτε ότι το λιμάνι αυτό ε, ε, βρίσκεται, ε, ε, είναι το, το κλειδί για τη σύνδεση με το Δούναβι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τη νέα στρατηγική και θα ήθελα ο εισηγητή να συμπεριλάβει τη σημασία ε, τη στρατηγική για το Δούναβι και τη ανάπτυξη του λιμανιού τη Κωνσταντ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Και πάλι μιλώ εκ μέρου του κυρίου Κούτα, ο οποίο σήμερα είναι δραστήριο και μου ανέθεσε να αναφερθώ σε όλα αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, βασικά, η πρωτοβουλία για μια κοινή στρατηγική για τον εύξηνο πόντο είναι πάρα πολύ θετική η πρωτοβουλία. Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, μεγάλο ενδιαφέρον και από πολιτική άποψη και από άλλες απόψεις. Δύο από τα ε, νέα κράτη-μέλη, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, βρίσκονται στον εύξηνο πόντο. Υπάρχουν και άλλες μερικές χώρες, η Ρωσία και τα λοιπά που είναι παραδουνάβιες χώρες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα στρατηγικής σημασίας. Ε, μας μα συνδέει άμεσα με την Τουρκία που είναι 7η και 5η αντίστοιχα σε εξαγωγέ και εισαγωγέ τη Ευρώπη. Ε, Επίση αναφέρω την Ρωσία που είναι βασικό εμπορικό εταίρο. Η Τουρκία και η Ρωσία λοιπόν ε, είναι απόλυτα ε, σημαντικέ χώρε στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική. Και αυτό ε, είναι ουσιώδε θέμα και πρέπει να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι με τη στρατηγική μα για, για τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την περιοχή. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε πολυάριθμα ζητήματα από κοινού. Εμπορικέ πτυχέ, αλλά και ευρύτερα θέματα όπως η διεύρυνση, η πολιτική γυτνίασης κτλ. Και όλα αυτά θα πρέπει να, να προχωρήσουν προς τον Νότιο Κάφκασο, Ευρωπαϊκή Προοπτική, Μολδαβίας και Ουκρανίας κτλ. Τελευταία παρατήρηση. Η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσε ε, να θεσμοθετηθεί ενδεχομένως σε ένα είδο ένωση που να περιέχει και μια κοινοβουλευτική διάσταση. Ε, ε, απλά το αναφέρω για να το σκεφτούμε. Και σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή για τον ε, επικοδομικό τρόπο με τον οποίο εξετάζει το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Δυστυχώ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι παρούσα. Ε, Μα ζήτησε συγγνώμη. Ε, Μάρτιν, θέλει να συνοψίσει σύντομα ή είσαι ικανοποιημένο με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Είναι αλήθεια ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βίνκλερ, δηλαδή πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και τους δρόμους της ενέργειας, τους νέους δρόμους που περνούν από όλη αυτή την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό στη γενικότερη προσέγγιση μας ως προς τη στρατηγική για τον εύξηνο πόντο. Ε, για τις συστάσεις ε, του συναδέλφου τώρα, να επιμείνουμε δηλαδή στη σημασία των λιμένων και κυρίως το λιμάνι της Κωνσταντσάς είναι ε, πραγματικά ε, σημαντικό θέμα, αλλά πάντοτε θα πρέπει να ε, συνδέουμε το θέμα αυτό με τις λοιπές ε, πρωτοβουλίες, όπως λέω και στην έκθεσή μου. Η στρατηγική για το Δούναβι, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν λιμένες στρατηγικής σημασίας. Υπάρχει και το λιμάνι του Βέρνερ, όχι μόνο της Κωνσταντσα. Ε, και που έχουν σημασία για τη διασύνδεση με τις οδικές και σιδηροδρομικές ε, μεταφορές. Ε, θα μπορούσα να αναφερθώ σε αυτό μέσα στην έκθεσή μου. Θα συμφωνήσω επίσης με τον κύριο Λάιχτε ότι χρειαζόμαστε ένα κατά τι ευρύτερο ε, πλαίσιο, πιο στοχευμένο από στρατηγική ε, πλευρά ε, για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες, όπως λόγου χάρη η εταιρική, ανατολική εταιρική σχέση και η πολιτική γειτονίας. Ευχαριστώ Μάρτιν. 5 Οκτωβρίου και πάλι η ημερομηνία για την υποβολή ε, τροπολογιών. Σημείο 11. Χορήγηση εγγύηση ΕΕ, ε, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύηση. Ε, Γουίλιαμ, ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε προεδρεύοντα θα έλεγα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι γιατί πλήττεται η νομιμότητά μου. Ε, κύριε Λάιφριντ και άλλοι συνάδελφοι, να σας πω ότι είναι και εγώ ερετός εκπρόσωπος είμαι ε, ε, και το κόμμα μου πήρε περισσότερες ψήφους στις ευρωπαϊκές εκλογές σε σχέση με το εργατικό κόμμα και τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές. Τι έκανα συντάσσοντας αυτή την έκθεση. Ε, απλούστευσα την φρασολογία που χρησιμοποιώ, διευκρίνησα το περιεχόμενο, εξορθολόγησα τις απαιτήσει ε, που προτείνει η έκθεση και έδωσα ιδιαίτερη έμφαση δεδομένης και της κατάστασης στο ότι ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να καταβάλουν υψηλότερους φόρους ε, δίνοντας ε, έμφαση στις αρχές της χρηστής ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης διέγραψα προτάσεις όπου αναφέρονταν αρχές ε, που μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους ε, στο ε, κόμμα μου και θα συμφωνήσω με τα σχολεία των συναδέλφων. Βίλιαμ, ευχαριστούμε. Ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ Ρόμπερτ και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. πρόσεξα ιδιαίτερα και διάβασα όλες τις τροπολογίες εντυπωσιακός αριθμό 45 που προτείνουν οι αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινώ λέγοντα ότι δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω με τι ε, αρχέ τη χρηστή ε, δημοσιονομική διαχείριση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Ε, αρχέ που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και που αντικατοπτρίζει και η διαγνωμοδότηση. Και νομίζω ότι οι νέε αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, θα πρέπει και αυτέ να εκφράζονται σε σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και στο Κοινοβούλιο, ενημέρωση, υποβολή έκθεση κτλ. Εγώ πιστεύω ότι η, τράπεζα, ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε για, ε, ε, για να υποστηρίζει ε, συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, με σημαντικές δυσκολίες μεν, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια συνεπή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν νομίζω ότι πολλές τροπολογίες για να χρησιμοποιήσω και τα ακριβή λόγια του διακεκριμένου συναδέλφου ε, δημιουργούν τρομερά προβλήματα, severely handicapped, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, π.χ. 22, 23 και 24, τροπολογίε τροπολογίες αυτές ε, που είναι διαγραφές. και που ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναλάβει τι εξωτερικέ τη δεσμεύσει και υποχρεώσει, κυρίω όσον αφορά τι ε, υποένταξη χώρε. Επίση, δεν συμφωνώ με το ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα πρέπει να έχει ε, του απαραίτητου πόρου ε, και σε ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπίσει τι νέε απαιτήσει. Για κάτι άλλο. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει στόχο να αφαιρέσει την Τουρκία από τον χώρο των επιλέξιμων χωρών. Από τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό και το κατά πόσον πόσο είναι υποψήφια χώρα η Τουρκία. Αλλά αν είναι υποψήφια χώρα, τότε μάλλον θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για ε, να συμπεριληφθεί στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν έχει το λόγο. Ναι, Ρόμπερτ. Με βοήθησε πολύ ο κύριος Βίγκλερ, γιατί με κάλυψε μεγάλο βαθμό. Και εγώ πιστεύω ότι ότι αυτή η πρόταση η οποία στοχεύει στον επανακαθορισμό των, ε, των προνομίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να, ε, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα στήρος χώρος δράσης της όπου δεν θα ε, εμπλέκεται σε μια στρατηγική ανάπτυξη συνεργασίας εν ώψη της διεύρυνσης και της προώθησης ορισμένων αξιών και προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι είναι κάτι το, πρέπει, ε, ε, το, το, ε, το οποίο συζητιέται ιδιαίτερα. Πρέπει να το συζητήσουμε, είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο. Επίσης, όσον αφορά την τροπολογία 44 για την αφαίρεση της Τουρκίας από τον κατάλογο του παρατήματος 2, εδώ νομίζω ότι η Τουρκία είναι μια χώρα με την οποία ήδη έχει συνάψει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χώρα υποψήφια για ένταξη. Εμεί είμαστε αυτοί που με μια τέτοια έκθεση θα αποφασίσουμε το αντίθετο. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Ο κ. Λάχιτφρεντ ναι, ήταν μάλλον προβλέψιμο αυτό. Νομίζω ότι η πρόταση είναι πολύ καλά εισαρπημένη, είναι πολύ θετική και πολλά θετικά στοιχεία περιέχει. Επί της αρχής είναι πολύ θετικό το ότι θα πρέπει να τονωθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να υποστηρίξει τους αναπτυξιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και επίσης οι δραστηριότητε, της σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα και σε ό,τι αφορά την, ε, τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν με κάποιο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, προκειμένου να υποστηριχθεί να υποστηριχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Ένωσης, να τονίσουμε δύο θέματα. Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η καταπολέμηση της ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη σε κάθε βήμα που θα κάνουμε για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΤΕΠ. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό θεωρώ. Ελπίζω κάτι να μας διδάξει αυτή η χρηματοοικονομική κρίση και ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε, ελπίζω, είναι ότι προκειμένου να προστατεύσουμε στο μέλλον καλύτερα τα δημοσιονομικά μας, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνονται δραστηριότητες στους φορολογικούς παραδείσους, όπως ονομάζονται. Και τέλος, ότι φυσικά θα πρέπει να γίνονται εκθέσεις ε, ελέγχου της διαφάνειας της ΕΤΕΠ. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω και εξ ονόματος μου, όχι εξ ονόματος του κυρίου Κούτας. Αν είχατε, κύριε Τάκμας, την ε, εντύπωση ότι σας έθιξα. Λυπάμαι, δεν εννοούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αμφισβητούμε την νομιμότητα των αποφάσεων που έχει λάβει το Κοινοβούλιο, γιατί και αυτό δεν είναι νομιμό με τη σειρά του. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Σαντό. Ε. Ευχαριστώ συχνά είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει του συναδέλφου Ντάρτμουντ γιατί αναζωογονούν τη συζήτηση και την καθιστούν πιο διασκεδαστική. Βέβαια όμω είναι πιο ενοχλητικά τα πράγματα όταν μεταφέρει τι ιδέε του μέσα σε εκθέσει. Σήμερα Έχουμε ε, ε, τρεις ε, εκθέσεις που αποσκοπούν στο να κατανομήσουμε καλύτερα τους τρόπους λειτουργίας του εμπορίου σε σχέση με τους κανόνες της κοινωνίας και τώρα έχουμε μια έκθεση με εντελώς αντίθετο περιεχόμενο, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να απεξαρτοποιηθεί από τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κλιματικά θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή είναι εντελώς αντίστροφο το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης σε σχέση με αυτό που προτείνουμε γιατί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη μελλοντική της λειτουργία. Εμείς ε, θα υποβάλουμε προφανώς τροπολογίες σε σχέση με αυτές τις προτάσεις και εξάλλου θα υποβάλουμε τροπολογίε και για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι θεωρούμε ότι προς το παρόν ε, ο τρόπος χειρισμού των κριτηρίων για τη χρηματοδότηση ε, δεν επαρκεί. Δείτε σήμερα η ΕΤΕ χρηματοδοτεί 9 δις ευρώ για, τις, για την πυρηνική ενέργεια και για τα ορυκτά καύσιμα και 6 δις, πολύ λιγότερο δηλαδή, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια παρά την συνένεση επίπεδο ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτή τη στιγμή σε περισσότερο οι ΕΤΕ στα κλιματικά θέματα. Εμείς ε, θα είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε τι σημαίνει αυτό να χρηματοδοτήσει η ΕΤΕ, δηλαδή την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι αν πρόκειται για τα βιοκαύσιμα, για τα μεγάλα φράγματα ή τη δέσμευση του άνθρακα, προφανέστατα εμείς ε, θα ταχθούμε κατά. Ευχαριστούμε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο, έκθεσης, το σχέδιο γνωμοδότησης του ε, και εμείς θέλουμε να απλουστευτεί το κείμενο όπως και ο εισηγητής. Επίσης ε, θέλετε να υπάρχει διαφάνεια, να ξέρουμε ποιος είναι υπόλογος, συμφωνούμε. Ακούσαμε και κάποια σχόλια από άλλα μέλη της Επιτροπής ε, και συμφωνούμε. Παραδείγματο χάρη τα μέσα για να υποστηρίξουμε την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κυρίως όταν μιλάμε για χρηματοδότηση προγραμμάτων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θέλουμε ε, να υποστηριχθούν τροπολογίες που υποβαθμίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα αυτό επίσης. Έχουμε επιφυλάξει σχετικά με την διαγραφή της Τουρκίας από τον κατώ Λέγω και την αναφορά του Καλίνιγκραντ σε παρένθεση Επίσης, ε, ποιο ήταν το πνεύμα της ε, πρότασής μας, ε, δηλαδή να αλλάξουν εξωτερικές δράσεις της ΕΤΕ ως προς τις κλιματικές αλλαγές, αυξάνοντας σταδιακά τον αναπτυξιακό ρόλο αυτής της τράπεζας. Οπότε και πάλι όλες αυτές οι τροπολογίες που προτείνουν το αντίθετο, μείωση δηλαδή υποβάθμιση του ρόλου ως προς τις κλιματικές αλλαγές, δεν μας βρουν σύμφωνους και θα συμφωνήσουμε και με τους ενδιασμούς του κυρίου Βίνκλερ για κάποιοι αρχές από τις αιτιολογικές σκέψεις ε, που διαγράφησαν αλλά συνιστούν σημαντικά στοιχεία, δηλαδή το ρόλο της τράπεζας, τη δυνατότητα που θα έχει να χρησιμοποιήσει περισσότερο τις εγγυήσει ε, ε, και επίσης τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, όλες αυτές οι λύσεις ε, αυξάνουν τις δυνατότητες ε, που έχει η ΕΤΕ να υποστηρίξει οι προγράμματα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε κάποιες τεχνικές διευκρινήσεις. Υπάρχουν και κάποια νομικά τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με κάποιες από τις τροπολογίες, αλλά μάλλον είναι θέμα της νομικής υπηρεσίας και όχι δικό μου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και... Ναι, με ακούτε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την πρόταση αυτή. Σε γενικέ γραμμέ, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση και τη σαφήνεια του κειμένου. Τονίζουμε τη σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση και την ενίσχυση της καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων. Αυτό ασφαλώς μας βρίσκει σύμφωνους, άλλωστε το κάνουμε ήδη και σήμερα. Και η σχετική υπηρεσία είναι πρωτοπόρος υπηρεσία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα συνεχίσουμε ωστόσο να τονίζουμε την πολιτική αυτή. Τώρα για κάποια από τα επιμέρους στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν για τις χώρες ε, που θα περιληφθούν. Δεν είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε ποιες θα είναι. Έχουμε πέντε επιπλέον χώρες και θα πρέπει να τονίσουμε ότι όπως αναφέρθηκε στην ενδιάμεση αναθεώρηση με την προσθήκη νέων χωρών κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουμε στο όριό μας, το το όριό μας πριν από το τέλος του 2013 θα είναι μάλλον περιορισμένο το πεδίο εφαρμογής μας στις νέες χώρες, ιδιαίτερα στη φάση της την της πρώτερη φάση της ε, εγκατάστασης και στην Ασία και στην ε, Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να ενισχυθούν οι σχέσεις αυτές αλλά και η υποστήριξη των πολιτικών μας και των αναπτυξιακών πολιτικών σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο μας ζητήσει κάτι τέτοιο. Τέλος, είναι σημαντικό για εμάς, ιδιαίτερα αν μας ζητηθούν πιο πολλές ε, δραστηριότητες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Ένωσης, να υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι, οι σωστοί πόροι η κατάλληλη χρηματοδότηση. Άρα η πρόταση να αφαιρεθεί η σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης και του τι ε, περιμένουμε από την τράπεζα θα πρέπει να ξαναεξεταστεί. Και ο λόγος και πάλι στο William. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρόκειται για συνεδρίαση της Επιτροπής και είναι πιο σημαντικό στις Επιτροπές να κοιτάμε στα σημεία επί των οποίων συμφωνούμε. βρήκαμε κάτι με τον οποίο συμφωνούμε τον κύριο Λάιχτφριντ. Τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει η Τράπεζα Επενδύσεων να μην παραμελεί το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και επίσης συμφωνώ σε ό,τι αφορά τα σχόλια που έγιναν για τη σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Να τονίσω όμως ότι η πολιτική στόχη σε πολλές περιπτώσεις είναι αντίθετη με την καλή, σωστή διαχείριση. Μπορεί να συνδυάσει κανείς και τα δύο, αλλά δύσκολα. Είμαστε πολιτικοί και πάντα θέλουμε να θέτουμε πολιτικούς στόχους. Είναι όμως δύσκολο να υπάρχουν πολιτικοί στόχοι, οι οποίοι συχνά είναι αντίθετοι με τις αρχές της ε, χρηστής διακυβέρνησης, διαχείρισης. Πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την χρηματοοικονομική κρίση όντως, και ο καθένα βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι η διαφάνεια είναι ωφέλιμη, προκειμένου να μην συμβεί ξανά το ίδιο. Και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που υπάρχει υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκ των ομιλητών ότι η ΕΤΕΠ θα πρέπει να διέπεται από απόλυτη διαφάνεια. Συμφωνώ με τα σχόλια της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη σαφήνεια, την οποία προσπάθησα να βάλω στο κείμενο και στις τροπολογίες. Και τέλος, αναφορικά με αυτά που είπε ο κύριος Ζαντό. Ασφαλώς και ανάμενα να υποβάλλετε τροπολογίες. Δεν φαντάστηκα ότι θα πρότεινα μια τέτοια έκθεση χωρίς τροπολογίες και να το πάω και παραπέρα. Θα με απογοητεύατε αν δεν υποβάλλατε τροπολογίε κύριε Ζαντό, και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Και να πω ότι πραγματικά ήταν αξιοζήλευτος ο επαγγελματισμός των όσων με βοήθησαν, ιδιαίτερα εκ μέρους της τράπεζας. Να δούμε τι θα επιζήσει μετά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γουίλιαμ, λέει ο Πρόεδρος. Σε συγχαίρω για την πρώτη σου γνωμοδότηση, για την πρώτη σου έκθεση. Ευχαριστούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και να περάσουμε στην ε, συνεδρίαση των ε, συντονιστών. 5 Οκτωβρίου, William. 5 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και τώρα να περάσουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Να παρακαλέσω όσοι δεν είναι συντονιστές να βγουν από την αίθουσα AUTHORWAVE